Good morning. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καθίστε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Καλώς ορίσατε. Αρχίζουμε τη σημερινή πρωινή συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Ε, αρχίζουμε την έγκριση μερίσιας διάταξης που έχετε μπροστά σας. Συμφωνείτε? Προχωρούμε. Ανακοινώσεις ε, του Προέδρου. Το γλωσσικό προφίλ είναι το γνωστό και ζητώ συγγνώμη που δεν έχουμε στη συγκεκριμένη συνεδρίαση διερμηνία στα μαλτέζικα, λετονικά και εγωιδελικά ιρλανδικά. Δυστυχώς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ε, όλες οι υπόλοιπες επίσημε γλώσσες παρέχονται. Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Προχωρούμε στην έγκριση ε, των ε, συστάσεων των συντονιστών έγινε μια πολύ εντατική συνεδρίαση των συντονιστών. Ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις, ε, τις οποίες και συνοψίζω. Για το ενημερωτικό σημείωμα αναφέρονται ε, εισηγητές ο κύριο Χόρχε Γουσαδέ για το Eurodac. Η κυρία Μπίργκετ Σίπελ, η εισηγήτρια ε, για τη σύσταση ε, για απόφαση του Συμβουλίου και όσοι αφορά τις διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Ηνωμένε Πολιτείες για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία και η κυρία Σίπελ πάντα και επίσης η συγκίτρια για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το ηλεκτρονικό έγκλημα ή το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Αν συμφωνείτε να εγκρίνουμε τις αποφάσεις των συντονιστών. Το λόγο έχει ζητήσει ο κύριος Μπουσαντέ. Έχετε το λόγο, είναι δικαστικό για ένα λεπτό. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όντως, ε, η το εγκλημα στον χωρο αν συμφωνειτε να εγκρινουμε τις αποφασεις των συντονιστων το λογο εχει ζητησει ο κυριος μπουσαντε εχετε το λογο ειναι δικαστικο για ενα λεπτο ναι ευχαριστω πολυ κυριε προεδρε οντως η ομαδα μας διαφωνεί με την πρόταση και τη σύσταση που ελήφθη από τους συντονιστές για την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει πρόταση μεταρρύθμισης για τη βελτίωση του συστήματος ε, Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Ανεβλήθη αυτή η απόφαση. Εμείς θεωρούμε ότι είναι κατεπίγουσα ε, έχει ελλείμματα, έχει προβλήματα, δεν γίνονται σεβαστά τα δικά συστήματα των κρατών μελών και ε, ε, χιλιάδες κλιματίες αλωνίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ε, ένταλμα ε, για να εξασφαλίσουμε τον κοινό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Τα στοιχεία της Eurostat ε, λένε ότι έχουν εκτελεστεί το 2016, που είναι το τελευταίο έτος που έχουμε στοιχεία, μόλις το 30% των ενταλμάτων σύλληψης. Δεν έχουμε χρόνο, ούτε μια εβδομάδα, ούτε ένα μήνα, πόσο μάλλον να περιμένουμε την καινούργια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τούτο εδώ το Κοινοβούλιο θα πρέπει να πάρει πρωτοβουλία για το θέμα αυτό και σύμφωνα με το άρθρο 214 του εσωτερικού κανονισμού προσβάλουμε προσβάλλουμε την απάντηση των συντονιστών και ζητούμε να ψηφιστεί εδώ στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ κύριε Μπούσαντε. Γνωρίζετε καταρχάς ότι η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης είναι κάτι το οποίο απασχολεί διάφορα ε, κόμματα και πολιτικές ομάδες. Εμείς δεν αποφασίσαμε απόρριψη, απλώς αναβολή της έγκρισης εκθέσεως πρωτοβουλίας ε, για τη λειτουργία και την ε, εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης. για οποιαδήποτε ενίσχυση ή τροποποίηση του εντάλματος. Η απόφαση λοιπόν των συντονιστών που εγκρίθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό μας ήταν να αναβληθεί η συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Ενταλμα και την αντίστοιχη έκθεση πρωτοβουλίας. Οπότε, Δεδομένου ότι η ομάδα σας, η η ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών ε, προβάλλει αντίρρηση στην αναβολή της απόφασης και ζητάει να ψηφιστεί, προτείνω το εξής. Το σημείωμα ε, που σας υποβλήθηκε από τους συντονιστές να εγκριθεί με εξαίρεση το συγκεκριμένο θέμα και να τεθεί σε ψηφοφορία αυτή η αναβολή της απόφασης για την έκθεση πρωτοβουλίας εν το χρόνο, στην επόμενη συνεδρίαση. Να το γνωρίζουν όλες οι πολιτικές ομάδες για να προσανατολιστούν και να ληφθεί η απόφαση. Και αυτή η συνεδρίαση κανονικά είναι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ ε, Δημοσίων Ελευθεριών, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 16 του μηνός στο Στρασβούργο. και θα ακούσουμε τον ε, απερχόμενο ε, επίτροπο, τον κύριο ε, Δημήτρη Αβραμόπουλο. Έχουμε συνεδρίαση στο Στρασβούργο στις 16 του μηνός τη Δευτέρα και προτείνω να μπει στην ημερήσια διάταξη ψηφοφορία για να το γνωρίζουν τα μέλη, να είναι παρόντα, να ψηφίσουν ανάλογα με τον προσανατολισμό και τις απόψεις της κάθε ομάδας. Εγγράφεται λοιπόν αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη της 16ης. Κύριε Μπουσαντέ. Κατανοώ ότι προεδρεύετε εσείς, αλλά διαφωνώ. Είμαστε όλοι ενήμεροι, συνεδριάζεται αυτή τη στιγμή κανονικά η Επιτροπή μας και μπορούμε να ψηφίσουμε. Ξέρω ότι εσείς ε, μπορείτε να αποφασίσετε, αλλά διαμαρτύρομαι. Εντάξει, δεν είναι παρόντα όλα τα μέλη της Επιτροπής και εγώ τι φταίω. Ούτε η πολιτική μου ομάδα φταίει, ούτε κανένας άλλος ε, από τα μέλη του Προεδρείου. Κοιτάξτε, Κανονικά θα πρέπει οποιαδήποτε ψηφοφορία να ανακοινώνεται εγκαίρως έτσι ώστε να, να ενημερώνουν ε, τα μέλη τους οι πολιτικές ομάδες και να έρχονται έτσι ώστε η ψηφοφορία να αντανακλά πιστά τις πλειοψηφίες στην Επιτροπή. Ευχαριστώ. Προχωρούμε λοιπόν. εγκρίνουμε τους υπόλοιπους ορισμούς εισηγητών και προχωρούμε στο πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ε, ξέρετε, είναι πολύ φορτωμένη, όπως πάντα η ημερήσια διάταξη. Αρχίζουμε με παρουσιάσεις. Η παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης 2018 σχετικά με την εφαρμογή του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θυμηθείτε ότι μαζί με τη συνθήκη της Λισαβόνας τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκέμβρη 2009 και ο χάρτης θεμελιδών δικαιωμάτων που έχει την ίδια ισχύ με τις συνθήκες. Το άρθρο 6 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει αυτά ε, και δίνει την ίδια ισχύ στο χάρτη των θεμελιδών δικαιωμάτων ε, που είναι πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης και ε, μπορεί κανείς να προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και υπάρχουν ήδη αποφάσεις πολλές που λέγουν ότι ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι δεσμευτικός για όλα τα κράτη-μέλη. Φυσικά και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Όταν πρόκειται για την εφαρμογή ή την υλοποίηση του ευρωπαϊκού δικαίου. Αυτό θα πρέπει να το γιορτάζουμε, να το παναγυρίζουμε, να το διατρανώνουμε προς τα έξω. Ε, και θα ακούσουμε την κυρία Μπάρμπαρα Νόλα, που είναι τμήματάρχη στη Γενική Διεύθυνση Τζά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά θα ακούσουμε τον Μάικλ Οφλάχερτη από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Και χαιρόμαστε που σας ε, βλέπουμε. Κύριε Οφλάχερτη, ξέρετε ότι ο Οργανισμός Θεμερινών Δικαιωμάτων εδρεύει στη Βιέννη. Αρχίζουμε λοιπόν με την παρουσίαση της κυρίας Μπάρμπαρα Νόλαν. Εξ όσων έχω καταλάβει, προσεχώς, σε διάφορα θεσμικά όργανα θα υπάρξουν συζητήσεις, συνεδριάσεις, πάνελ, ε, στρογγυλές τράπεζες για να ε, εκτιμήσουν σωστά ε, την εκτέλεση αυτή τη δεκαετία του Χάρτη Θεμελιδών Δικαιωμάτων. Είναι μια, η επέτειος των 10 ετών και τις επόμενες εβδομάδες θα συμμετέχουμε και εμείς σε αυτές τις συζητήσεις. Πραγματικά είναι ένα γεγονός άξιο σημείο του και θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, διότι ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Θεμελιδών Δικαιωμάτων ήταν άλμα για ιδιαίτερα ε, ε, ε, για την εδραίωση της ίδιας της έννοιας της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη. Κυρία Νόλαν, έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και καλημέρα σε όλους και στους νέους βουλευτές και σε εκείνους που γνωρίζω από το παρελθόν και όπω τα ξέρετε ορισμένοι από εσά, παρακολουθώντα τη θέση σε ισχύ τη Χάρτα των Θεμελιδών Δικαιωμάτων πριν από μία δεκαετία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια στρατηγική για τη Χάρτα. Που μεταξύ άλλων αναλαμβάνει τη δέσμευση να υποβάλλεται ετήσια έκθεση για την εφαρμογή αυτή από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη. Η ενάτη λοιπόν έκθεση για το 2018 υιοθετήθηκε τον Ιούνιο φέτος και αποτελείται από ένα σύντομο έγγραφο ε, εν είδη ανακοίνωσης καθώς και μια ε, λεπτομερέστερη υπηρεσιακή παρουσίαση. Είναι μια επισκόπηση για το πώς ε, εφαρμόστηκε η χάρτα το 2018. Το 2018 προφανώς πρέπει να ολοκληρωθεί για να μπορέσει κανείς να γράψει γι' αυτό. Η φετινή βέβαια χρονιά είναι εξίσου σημαντική, διότι γιορτάζουμε την 10 επέτειο από την θέση σε ισχύ της χάρτας και θα δείτε ότι η έκθεση εστιάζει και σε αυτό το επίπεδο του εορτασμού καθώς και το κατά πόσον ε, έγινε η ανακοίνωσή μας για την ευαισθητοποίηση περί χάρτας αντιληπτή από τον Ιούνιο όταν δημοσιεύτηκε. Λίγο απογοητευτικά τα αποτελέσματα. Πάντως στη δεκαετία αυτή τη βλέπουμε ότι η αντίληψη για τα θεμελιώδη δικαιώματα κάπως ε, βελτιώθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση περιγράφει πρωτοβουλίες που προωθούν απευθείας τα θεμελιώδη δικαιώματα και σε τομείς όπου τα δικαιώματα αυτά παραμένουν ε, προτεραιότητα όπως απαιτεί η Στατηγική της Επιτροπής. Η έκθεση του 2018 επικεντρώνεται κυρίως στα νέα δικαιώματα για τη δικαιοσύνη, καθώς και το Ταμείο για τις Αξίες. Αυτά παρέχουν περαιτέρω στήριξη για του υπερασπιστέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τι οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών που ενεργοποιούνται στον τομέα τη προστασία των δικαιωμάτων. Ε, πρωτοβουλία για του καταγγέλλοντε, την οποία θα γνωρίζετε περισσότεροι. Και Μάλλον θα τεθεί σε ισχύ αργότερα φέτος αυτή. Το πακέτο για τι εκλογέ αυτό είχε παρουσιαστεί πριν τι ευρωεκλογέ, καθώ και το σχετικό συνέδριο για τη δημοκρατία, ε, που οργανώθηκε στα τέλη της περσινής χρονιάς υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου Τίμερμαντς. Επίσης υπογραμμίζεται η διαρκής προσπάθεια να καταπολεμηθούν οι εκφράσεις μίσους ε, στο διαδίκτυο και να βελτιωθεί και η διαδικασία ένταξη των Ρωμά. Το πρώτο σκέλο είναι να μιλήσω για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων και το, την παρακολούθηση τη εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σε σύγκριση με προηγούμενες εκθέσεις βλέπουμε ότι ένα μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού δικαίου και των πολιτικών προωθούν απευθεία τα ίδια στοιχεία με την ε, χάρτα για την προστασία των θυμάτων, την ε, ε, νομική προστασία, την ισορροπία επαγγελματικού και γενικού βίου και την ευθυγράμμιση της διάστασης των φύλων. Η χάρτα δεν μιλάει απευθεία για, ε, για το πώς πρέπει να αναλυθούν δράσεις για την προστασία των δικαιωμάτων. Έχουμε όμως κάποιες πρωτοβουλίες με την Επιτροπή ε, με κατευθυντήριες γραμμές και κατάρτιση συναδέλφων από άλλες γενικές διευθύνσεις για να μπορέσουν να δουν κατά πόσο οι δικές τους πρωτοβουλίες συνάδουν με τους στόχους της χάρτας των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο να αναπτύσσουν καλά αντανακλαστικά οι συνάδελφοι αυτοί, τα οποία ανταποκρίνονται και στη στου στόχου τη δική μα υπηρεσία, όπου ελέγχουμε όλα τα σχέδια των δράσεων που οργανώνονται. Αυτή η διαδικασία παρακολούθηση επιθεώρησης είναι πολύ σημαντική ω συνοδευτικό τη νομοθετική διαδικασία. Διότι πριν φτάσουν σε εμά οι προτάσει σα, έχουμε κάνει αυτή τη δουλειά. Οπότε, όταν κι εσεί λάβετε τι προτάσει, ω Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, έχετε ένα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσετε. Να κοιτάξετε κατά πόσον έχουμε κάνει σωστά τη δουλειά μα δηλαδή. Και πράγματι, μπορείτε να τοποθετηθείτε για το θέμα τη συμμόρφωση με τι απαιτήσει για τα θεμελιώδη δικαιώματα και σε σχέση με κάθε νομοθετικό ντοσχέ που πριν από το Κοινοβούλιο. Υπάρχει λοιπόν μια αρχή γενική που διέπει όλη τη δουλειά για να δούμε κατά πόσον τα θεμελιώδη δικαιώματα γίνονται σεβαστά ή όχι. Επίση, η Επιτροπή σα συμβάλλει στην καλλιέργεια μια καλή νοοτροπία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και γενικότερα το σεβασμό του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώ και τη συμπερίληψή του σε πολλέ νομοθετικέ εκθέσει, ιδέε πρωτοβουλία εκθέσει ή προφορικέ ερωτήσει. Πώ παρακολουθούμε την κατάσταση στα κράτη-μέλη τώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει θεματοφύλακα των συνθήκων. Η χάρτα πρέπει να γίνεται πλήρω σεβαστή από τα κράτη-μέλη όταν εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο και αυτό είναι κέρια σημασία. Η χάρτα μπορεί να εφαρμόζεται μόνο όταν τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν και το ευρωπαϊκό δίκαιο ταυτόχρονα. Η Επιτροπή παρακολουθεί την κατάσταση επιτόπου και κινούμε επί παραβάσει διαδικασίες όταν βλέπουμε ότι η συμμόρφωση είναι πλημελή. Επίσης, δεν χρειάζεται να το θυμίσω φαντάζομαι, αλλά καλό είναι να το πω, ότι έχουμε ξεκινήσει πολλές διαδικασίες ε, επί παραβάση σε σχέση με τα θέματα των αξιών στην Ουγγαρία, ιδίως για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, την ε, ελευθερία των ακαδημαϊκών και το δικαίωμα στο άσυλο καθώς και την ε, υποστήριξη των ετών άσυλων. Οι περισσότερε από αυτέ τι διαδικασίε εκκρεμούν αυτή τη στιγμή, δεν έχουν εκδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και πρόσφατα έστειλε μια επίσημη επιστολή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ την Ουγγαρία για την παροχή τροφίμων σε όσους αναμένουν την επιστροφή τους τον επαναπατρισμό τους και βρίσκονται σε περιοχές διέλευσης ε, της Ουγγαρίας, ιδίω κοντά στα σύνορα με τη Σερβία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση εκκίνησε διαδικασία κατά της Πολωνίας ε, για το πρωτογενές δίκαιο, το δίκαιο για τα πρωτοβάθμια δικαστήρια και το τι γίνεται με το διορισμό των δικαστών, των δικαστικών λειτουργών. Η δεύτερη υπόθεση εκκρεμεί ε, και αναμένουμε απόφαση το φθινόπωρο. Βάσει τη νομολογία επίση η έκθεση δείχνει ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή διαρκώ παραπέμπει στη χάρτα στα κείμενα των αποφάσεών του. Δηλαδή αρχίζει να είναι περισσότερο προβεβλημένη και αντίληπτη η λειτουργία της χάρτας. Επικαλείται τα της χάρτας στο δικαστήριο στις αποφάσεις του, ιδίω ως προς τους αριθμούς. 356 υποθέσεις το 2018 σε σύγκριση με μόνο 27 το 2010. Ήταν περιπτώσεις που αναφέρθηκε η χάρτα. Να θυμόμαστε ότι η χάρτα είναι σχετικά νέο εργαλείο, νεαρό στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Χρειάζεται λοιπόν χρόνος μέχρι να μαθευτεί και οι κύριοι πρωταγωνιστές να ξέρουν ότι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Πάντως βλέπουμε ότι αρχίζει να δημιουργείται πρόσφορο έδαφος. Επίσης, ε, πολλές φορές και οι δικαστικοί των κρατών μελών ε, ζητούν ε, βοήθεια στην εκδίκαση υποθέσεων με 84 προδικαστικά ερωτήματα του 2018 και 19 μόλις το 2010. Θα βρείτε τα αριθμητικά στοιχεία και στην έκθεση. Το γεγονός ότι η χάραξη τη δικαστική πολιτική από του από δικαστέ γίνεται πλέον με ευρεία χρήση τη χάρτα είναι σημαντικό και θα επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων στην φάση της επιβολής της αλυσίδας, για να το πω έτσι, της εφαρμογής του νόμου. Παρόλα αυτά, η χάρτα δεν αξιοποιείται στο πλήρες δυναμικό της, καθώς και η ευαισθητοποίηση που μπορεί να υπάρξει μεταξύ των πολιτών δεν είναι μεγάλη. Αυτό είναι κάτι που πρέπει όλοι μαζί να το επιδιώξουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, όπου προεδρεύει ο Μάικλ, ή μάλλον για τον οποίο θα σας μιλήσω ο Μάικλ, στην έκθεσή του αναφέρει την έλλειψη εθνικών πολιτικών για την προώθηση της χάρτας, την ευαισθητοποίηση, το Ευρωβαρόμετρο που ανέφερα Στη μελέτη του από τι αρχέ τη Χρονιά, δείχνει ότι παρόλο που η κατάσταση έχει κάπω βελτιωθεί από το 2012, δείχνει ότι 4 στους 10 πολίτε μόνον γνωρίζουν την ύπαρξη τη χάρτα. και μόνο ένα στου 10 ξέρει τι ακριβώ λέει. Ένα, 6 στου 10 λένε ότι θα ήθελαν περισσότερε πληροφορίε για τα δικαιώματα που παρέχει η χάρτα και θέλουν να ξέρουν και πώ μπορούν να αξιολογούν αν παραβιάζονται τα δικαιώματά του. Έχουμε λοιπόν τεράστια δουλειά μπροστά μα για να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τα θέματα τη χάρτα, ιδίω σε εθνικό επίπεδο. Έχουμε συλλογική ευθύνη να ενημερώσουμε Και η χάρτα πραγματικά μπορεί να φέρει διαφορά στην ζωή των ανθρώπων μόνο αν γνωρίζουν τα δικαιώματά του, αν γνωρίζουν ότι τα δικαιώματά του παραβιάζονται, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με τρόπο ιδιαίτερα ε, προσεκτικό, ώστε να μην εφαρμόζεται ανεξαρτήτως των ε, συνθήκων. Μην ε, δημιουργήσουμε μεγάλες προσδοκίες και ευσεβείς πόθους ότι η χάρτα μπορεί να λύσει όλων τα προβλήματα. Έχει και αυτή τα ωριά της. Το γνωρίζετε εσείς βέβαια ως ευρωβουλευτές. Τα πολιτικά δικαιώματα, τα δικαιώματα της κοινωνίας των πολιτών δηλαδή, των ακτιβιστών είναι ύψης της σημασίας για την ευαισθητοποίηση, με τους φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους ε, φορείς που ασχολούνται με τα θέματα ισότητας πρέπει να συνεργαστούμε, καθώς και με τους δικηγόρου που ασχολούνται με τα θέματα ε, αυτά, καθώς και τους δικαστικούς λειτουργούς. Εκεί χρειάζεται κατάρτιση και εκπαίδευση για τα δικαιώματα της χαρτάς, για τις αρχές και τις αξίες. Μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε στην εκπαίδευση των νομικών και των δικαστικών λειτουργών και θα έχουμε περισσότερες δυνατότητες βάσει του νέου ταμείου για να προβλέψουμε περισσότερη εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι δικηγόροι και οι προεσπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να έχουν περισσότερες πληροφορίες στα χέρια τους για τη χάρτα, καθώς βρίσκονται σε άμεση επαφή με τους πολίτες Εκείνοι μπορούν να εξηγήσουν καλύτερα ποια ακριβώς είναι τα δικαιώματα και με το e-justice, την ηλεκτρονική δικαιοσύνη, μπορούμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες γενικές για το τι περιλαμβάνει η χάρτα. Εν είδη συμπεράσματο, καλύτερη χρήση και ευαισθητοποίηση της, για τη χάρτα θα είναι στο επίκεντρο τη εκδήλωση που θα οργανώσουμε επί Φιλανδική Προεδρία με τον Οργανισμό για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στι 12 Νοεμβρίου εδώ στι Βρυξέλλε. Θα είναι μια τέλεια ευκαιρία για να γιορτάσουμε τη 10η επέτειο τη χάρτα. Ένα νομικό δεσμευτικό εργαλείο και να ε, σκεφτούμε πώς ε, με τη συνεργασία όλων των φορέων της επιβολής ε, του νόμου, ιδίω με τις εθνικές αρχές, τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μπορούμε να αναπτύξουμε τη συνεργασία μα περαιτέρω για να εφαρμοστεί καλύτερα χάρτα. Χαίρομαι που θα έρθει και ο πρόεδρο τη Επιτροπή σα ε, στην εκδήλωση αυτή και όλοι μαζί θα μπορέσουμε να εξετάσουμε το πόρισμα και να ε, προωθήσουμε τα αποτελέσματά του. Ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε που συνεχώς θυμίζω πόσο σημαντικό είναι να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Το ξέρουν τα μέλη της Επιτροπής, αλλά για όσους είναι εδώ καινούργοι, θα αντιληφθείτε γρήγορα ότι είμαστε από τους πιο πολύ άσχολους ε, στο Κοινοβούλιο. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο φόρτο εργασία. Και συστηματικά έχουμε πολύ φορτωμένες ατζέντε. Ο Επίτροπος King θα έρθει στις 9.45. Και είναι πολλοί οι συνάδελφοι που έχουν ζητήσει το λόγο. Θυμίζω λοιπόν τη σημασία του να σεβαστείτε το χρονικό περιθώριο. Δέκα λεπτά παρουσίαση θα έχουμε και από το Μάικλ O'Flaherty. όλοι οι οργανισμοί ε, που ασχολούνται με τα θέματα αυτά έχουν έρθει στην Επιτροπή Λίμπη και μας έχουν μιλήσει. Ξέρουμε τη δουλειά του Οργανισμού Θεμελιωδίου Δικαιωμάτων. Έχουμε εξετάσει κάθε έκθεσή τους. Διότι πραγματικά έχουν μια συνολική επισκόπηση του πώς εφαρμόζονται τα δικαιώματα του, αν υπάρχει διακριτική μεταχείριση, τις απειλές που ανακύπτουν ε, στο σκηνικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Γι' αυτό, Μάικλ Φλάχερτη, στο επόμενο δεκάλεπτο, πες τόσο πιο γρήγορα μπορείς παρακαλώ, για να ακούσουμε και πολλούς συναδέλφους και να ολοκληρώσουμε γύρω σε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ευχαριστώ. Ε, πολύ κύριε Πρόεδρε. Λαμβάνω υπόψη την προειδοποίηση για τον χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό ημέρα σας. Είναι πλέον ε, μόνιμη μας πρακτική να σας υποβάλω την ετήσια μας έκθεση, αλλά πέρα από αυτό θα, ήθελα να σας παροτρύνω να χρησιμοποιήσετε αυτή την έκθεση και το περιεχόμενό της, που είναι πολύ χρήσιμο για τη δική σας σημαντική εργασία. Ε, δεν ήθιστε αυτό, αλλά εδώ έχουμε μια έκθεση όχι τόσο των υπηρεσιών, αλλά του διοικητικού μας συμβουλίου που υιοθετεί ετησίως αυτήν την έκθεση. Η έκθεση του 2019 περιλαμβάνει το περιεχόμενο που αφορά το 2018. Είναι δύσκολο τώρα κανείς να ε, διαλέξει ε, κάποια θέματα μόνο. Θα ήθελα λοιπόν αυθαίρετα να σας αναφέρω πέντε κοινότητες που κινδυνεύουν στην Ευρώπη και μετά κάποια ενθαρρυντικά μηνύματα. Πρώτη κοινότητα είναι οι Εβραίοι. Στη, Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα αντισημιτισμού στην Ευρώπη και μάλιστα η κατάσταση έχει ως εξής. Σημαντικό σημαντικός αριθμός των Εβραίων αδελφών μας ε, εξετάζουν τα δεχόμενα να καταλήψουν την Ευρώπη λόγω του αντισημιτισμού. Εμείς καλωσορίζουμε την αντίδραση σε όλα τα θεσμικά όργανα και στην Κομισιόν και σε αυτό το εδώ το Κοινοβούλιο που ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Δεύτερη κοινότητα που κινδυνεύει είναι οι μουσουλμάνοι ιδιαίτερα οι μετανάστες μουσουλμάνοι. Και εδώ βλέπουμε πάρα πολύ ανησυχητικά προβλήματα μίσους ε, προς εκείνους ε, και ε, συστηματικές διακρίσεις. Και πάλι σε ανταπόκριση αυτής της πολύ ανησυχητικής κατάστασης συγκεντρώσαμε στοιχεία από τις έρευνές μας και μετά από αίτημα της Κομισιόν έχουμε δημιουργήσει, δημιουργήσει μάλλον μια βάση δεδομένων για περιστατικά κατά των μουσουλμάνων και συντηρείται αυτή η βάση ε, μονίμως. Η τρίτη κοινότητα που ε, κινδυνεύει είναι η Ρωμά. Είναι η μεγαλύτερη μειονότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 6 εκατομμύρια κόσμο περίπου και όπως όλοι γνωρίζετε πολύ καλά υπάρχουν εντυπωσιακά στοιχεία ε, περιθωριοποίηση ε, και ανισότητας. Ε, η στήριξη για τη θεμελιώδη δικαιώματα των Ρωμά παραμένει προτεραιότητα και για τα επόμενα χρόνια για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Έχουμε λοιπόν όχι μόνο δεδομένα αλλά και τα σχήματα αντιθυγκανισμού, δηλαδή μίσος κατά των ανθρώπων αυτών ακριβώς επειδή είναι Ρωμά. Η τρέταρτη κοινότητα είναι οι μετανάστες. Ε, Εξεκολουθεί αυτή, αυτός ο τομέας να είναι τομέας όπου εστιάζει την προσοχή ο οργανισμός μας. Δεν χρειάζεται να σας πω πολλά πράγματα για την κατάσταση. Γνωρίζετε πολύ καλά τι συμβαίνει. Από το 18 μέχρι και το 19 μεγάλο μας προβληματισμός ήταν η κατάσταση στη Μεσόγειο και ιδιαίτερα τα περιστατικά πνιγμών στην θάλασσα. Το 2018 έξι άνθρωποι την ημέρα πνίγονταν και συνεχίστηκε αυτή ε, η κατάσταση μέχρι τους τελευταίους μήνες. Ανησυχούμε πάρα πολύ για ε, την συσχέτιση της, ε, μάλλον για το σχετικό επίσης περιστατικό που είναι η ποινικοποίηση των, της διάσωσης. Η τέταρτη κοινότητα είμαστε εμείς, ο γευρύτερος πληθυσμός. Για το 2018 συνειδητοποιήσαμε και καταλάβαμε πόσο πολύ η ιδιωτική μας ζωή κινδυνεύει και υποβαθμίζεται στο πλαίσιο της ψηφιακής ε, ζωής. Ε, γι' αυτό και ε, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για προστασία των προσωπικών μας στοιχεία όσον αφορά τη λειτουργία του ίντερνετ. Πέντε κοινότητες λοιπόν, πέντε ομάδες ανθρώπων για τους οποίους ανησυχούμε ε, το 2018, το ίδιο συνεχίζεται και το 2019. Αλλά δεν είναι μόνο η ανησυχία και η αρνητικότητα. Θα σας ε, πω και πέντε σημαντικούς τομείς ε, όπου έχουμε ενδείξει ελπίδα το 2018. Το 2018 είδαμε πολύ σημαντικές σημαντικά νομοθετήματα που υιοθετήθηκαν ή που είναι υπό εξέλιξη για να καλύψουν αυτές μας τις ανησυχίες. Βεβαίως, η σημαντικότερη από αυτές, το σημαντικότερο το νομοθέτημα ήταν το GDPR. Έχουμε μάλιστα δημοσιεύσει ένα εγχειρίδιο ώστε στην πράξη να διευκολυνθούν όσοι πρέπει να εφαρμόσουν αυτή τη σημαντική και περίπλοκη νομοθεσία. Είδαμε επίσης ε, τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων να στηρίζεται περισσότερο και πολλά άλλα νομοθετήματα ενισχύθηκαν από την άποψη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μάλιστα χάρη στην εργασία της δικής σας Επιτροπή που συχνά ε, συμφωνεί με τι αναλύσεις που κάνουμε εμεί, α πούμε, στην κανονισμό αιτία, αλλά και όσον αφορά τον εσωτερικό κανονισμό μας. Ε, επίσης είδαμε ε, θετικά στοιχεία ε, στον τομέα της καλής πρακτικής σε εθνικό επίπεδο. Είδαμε ότι κάποιες χώρες τα καταφέρνουν σωστά και πρέπει να τα καταφέρουμε καλύτερα να γνωστοποιήσουμε αυτές τις καλές πρακτικές. Στην έκθεση που έχετε μπροστά σας έχουμε 30 παραδείγματα καλής πρακτικής σε εθνικό επίπεδο που θα έπρεπε να είναι περισσότερο γνωστά. Σας δίνω ένα παράδειγμα δημοσιεύσαμε μια έκθεση του 18 για τις καλές πρακτικές για την αποϊδρυματοποίηση των ανθρώπων με, με ειδικέ ανάγκες ε, και ο τέταρτος τομέας με θετικά στοιχεία είναι η νέα προσοχή που δίδεται όχι μόνο στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά στην αρχιτεκτονική που προστατεύει ενάντια σε τέτοιε καταπατήσει. Α πούμε, η Κομισιόν δημοσίευσε σημαντικέ συστάσει για να ενισχύσει το ρόλο των σωμάτων ε, που προστατεύουν την ισότητα. Για παράδειγμα, το 2018 πάλι είδαμε να εστιάζεται περισσότερο η προσοχή στη στήριξη τη κοινωνία των πολιτών. Αναγνώρισε ότι σε πολλά μέρη είναι υποποίηση και ότι χρειάζεται συστηματική ανταπόκριση από πλευρά των των ευρωπαϊκών θεσμών και ευρύτερα. Το 2018 ήταν σημαντικό γιατί δόθηκαν απαντήσει και πρωτοβουλίε και από πλευρά εδώ του Ευρωκοινοβουλίου για την ενίσχυση του κράτου δικαίου. Σε ένα, άλλο άλλος που μα δίνει θετικά στοιχεία για από το 2018 είναι τέταρτος από το, το τέταρτο από τα πέντε μου θετικά στοιχεία είναι η προσοχή στο χάρτη. Η Μπάρμπαρα Νόλαν είπε πολλά για το χάρτη ε, εγώ λίγα έχω να προσθέσω, αλλά να ε, προσθέσω μία ε, προσωπική παρατήρηση. δεν είναι τόσο η καταπάτηση του χάρτη, αλλά όσο η, η αγνόηση αυτού. Κανένας δεν έχει ιδέα για την Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 58 όταν φτιάχτηκε η Ένωση. Δηλαδή, ο κόσμος δεν ξέρει γι' αυτά. Πρέπει αυτό ε, που πρέπει να μας ενθαρρύνει και μέσα από πρωτοβουλίες φέτο προσπαθούμε να αναπτύξουμε εργαλεία ε, ώστε εσείς και τα κράτη να μπορέσετε να εφαρμόσετε το χάρτη, πότε εφαρμόζετε, πότε όχι. εμεί ερευνούμε επίση ε, μάλλον επενδύουμε σε μια εκδήλωση τον Νοεμβρίου ε, και σας ενθαρρύνουμε εσάς ως ΛΥΜΠΕ να αναλάβετε πρωτοβουλίες στις τελευταίες εβδομάδες αυτού του επαιτειακού έτους ώστε να δώσετε αυτή την όθεση στο πνεύμα ε, στο οποίο μίλησε η Μπάρμπαρα. Το τελευταίο εθαρρυντικό στοιχείο ήταν ότι επιτέλους η προσοχή που δίνεται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης ε, ε, και πώς αυτοί εφαρμόζονται εντός της Ένωσης ήταν σημαντική. Ήταν χώρια υπόθεση μέχρι πρόσφατα. Ενώ τώρα ε, παίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την εμπέδωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αρχών σε όλα τα θέματα τα αναπτυξιακά που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνίες. Και γι' αυτό το λόγο το θεματικό μας ε, κεφάλαιο της έκθεσης που έχετε εδώ μπροστά σας από, ε, τον οργανισμό μας αφορά την προώθηση των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης εντός της Ένωσης. Γι' αυτό κύριε Πρόεδρε, ε, αυτά έχω να σας πω. δεν εκφράζουμε βαρές και ήταν σκληρή χρονιά το 2018, αλλά είδαμε και κάποιες ελπίδες, κάποιες ακτίδες φωτός, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ και επειδή τηρήσατε το χρόνο σας και για την εξαιρετική εισήγηση, τις εξαιρετικές εισηγήσεις από την κυρία Νόλαν και εσάς. Είναι προφανές ότι ο Επίτροπος Κίνγκ θα χρειαστεί να περιμένει. Αλλά, αλλά μην περιμένει και πάρα πολύ. Είναι θέμα ευγένειας. Όσοι ήθιστε έχουμε ένα μεγάλο κατάλογο. 15 συναδέλφων που ζήτησαν το λόγο. Παρακαλώ λοιπόν ένα λεπτό έκαστος για να έχουμε και λίγα λεπτά για να ακούσουμε απαντήσεις. Διαφορετικά θα σας δώσω σε ορισμένου το λόγο και οι υπόλοιποι πείτε τα γραπτά. Εγώ πάντα προσπαθώ ωστόσο να σας ακούσω όλους. Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος. Αν κρατήσετε το χρόνο που σας δίνω, οκ. Αλλά αν όχι, θα είναι δύσκολα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Δεν έχουμε συγκεκριμένη σειρά. Ε, αρχίζουμε με την κυρία Σίπελ. Ένα λεπτό. Έκαστος. Κυρία Ιντεβέλντε, σας έχω γράψει και εσάς τον κατάλογο, μην βιάζεστε. Αλλά παρακαλώ ένα λεπτό μόνο να μιλήσετε. Λοιπόν, κυρία Σίπελ, εσείς πρώτη. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Είχαμε πολλές καλές ε, συζητήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις απειλές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω σε ένα σημείο που είναι η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη που ε, συνεχώς αυξάνει σημασία και τώρα σκέφτεται τίποτα Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ο ΟΘΑ, Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, για να προστατεύουμε τη ζωή μας. Παράδειγμα, η αναγνώριση προσώπου δεν χρησιμοποιείται μόνο στην επιβολή του νόμου, αλλά σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Τι λέτε, είμαστε προετοιμασμένοι. Η κυρία Νετφέλτ, δεν νομίζω να μπορώ να είμαι τόσο σύντομη. Ποιο είναι το πρόβλημα. Παίρνουμε αιτήσει εκθέσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οπλισμένη ε, με πολλές νομοθεσίες, συμβάσεις κτλ. Και από νομικής πλευράς έχουμε το καλύτερο σύστημα στον κόσμο. Το πρόβλημα είναι η επιβολή και η εφαρμογή, η οποία είναι πολύ ασθενής. Και είναι πολιτικό το πρόβλημα αυτό. Διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποτίθεται ότι υλοποιεί και εφαρμόζει, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φοβάται ουσιαστικά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πόσο ανεξάρτητη και πόσο ε, θαραλέα θα αποδειχτεί η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντως μέχρι τώρα δεν είναι ενθαρρυντικά τα σημάδια. Τούτη εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τολμήσει να ορθώσει το ανάστημά της απέναντι στα κράτη-μέλη. Ε, συνήθως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αφήνει σε μεμονωμένους πολίτες που είναι πρόθυμοι να μπουν σε αυτή τη δικαστική μάχη ε, για χρόνια αλλά αυτό που κάναμε εμείς για τον προϋπολογισμό βασικά το όπνιξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ μπορείτε να διαβιβάσετε αυτά σε πολιτικό επίπεδο. Η κυρία Στρίκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους δύο μιλητές για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις. Για την κυρία Νόλαν, υπάρχουν τρόποι κατά την άποψή σας να βελτιωθεί η διάσταση της διαφάνειας περί συμμόρφωσης με την χάρτα Πώ τα λαμβάνετε υπόψη στι μελέτε αντικτύπου και τι εκθέσει υλοποίηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνώ με την κυρία Ιντβελτ ότι η απτή η πραγματική υλοποίηση είναι εκεί που υπάρχουν τα πραγματικά προβλήματα. Τι τρόποι λοιπόν υπάρχουν να έχουμε πρακτικότερε κατευθυντήριε γραμμέ για του ε, υπευθύνου λήψη αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο και το πώ να εφαρμόζουν τη χάρτα, λόγω χάρη το άρθρο 24, το Βέλτε στο συμφέρον. Ε, του παιδιού που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη έχει ερμηνευτεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Επίσης, για την εξωτερική εφαρμογή εκτό εκτός επικράτειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Σουφλάχερτη ήδη ανέφερε τις διάφορες επιχειρήσεις εμ, διάσωσης στη Μεσόγειο και υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί που λειτουργούν εκτός Ένωσης. Πώς ε, διασφαλίζουμε και την συμμόρφωση με την χάρτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι έχουμε περάσει σε μια νέα φάση της πολιτικής. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε εξελίξεις που έχουν αλλάξει τελείως το διεθνές προσκήνιο και μιλάω για το Brexit, τις Αμερικανικές εκλογές το 2016 και τις πρόσφατες ε, εξελίξεις ε, στην Ευρώπη. Βλέπουμε πώς έχει αλλάξει η παραδοσιακή προεκλογική στατεία όπως τη γνωρίζαμε και ο τρόπος να κάνει κανείς πολιτική. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε τα εργαλεία ανάλυσης και επικοινωνίας που διαθέτουμε. Μέσω από την ψηφιοποίηση έχουν αλλάξει τελείω και επηρεάζονται πολλές φορές και τα εκλογικά αποτελέσματα. Αυτά που μας παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θετικά αποτελέσματα. Όμως υπάρχουν και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Δεν πρέπει να κάνουμε κάτι και για αυτές για να προστατεύσουμε τις μεγάλες δημοκρατικές αξίες δεν πρέπει να υπάρχει ένας μεγάλος ε, δημόσιος χώρος για διάλογο δημοκρατικό που να μπορούν να συμμετέχουν όλοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να καταπολεμήσει την ε, παραπληροφόρηση. Χωρί όμω αυτό να γίνει ένα εργαλείο λογοκρισία. Πώς μπορούμε να αναχαιτήσουμε αυτό το φαινόμενο στην πράξη προστατεύοντα το ίδιο το πνεύμα τη δημοκρατία. Απλώ να σα θυμίσω ότι ο επίτροπο King έρχεται σε λίγα λεπτά. Είναι το δεύτερο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Κυρία Γιάροκα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα κι εγώ να ακουστεί, να κάνω τη φωνή μου να ακουστεί, για τα δικαιώματα των Ρωμά. Ε, σωστά το είπατε. Και των παιδιών κυρίως. Στην Ευρώπη υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά που δεν μπορούν να πάνε σχολείο. Πριν έρθω εδώ σήμερα, φρόντισα να σας μεταδοθεί ένα βίντεο για να δείτε τι γίνεται με τα δικαιώματα των παιδιών σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για τα κράτη-μέλη να τα εφαρμόζουν όσα προβλέπουν τα ευρωπαϊκά νομοθετήματα και κανένα ε, δεν παρακολουθεί πώ εφαρμόζονται. Μιλάμε για δικαιώματα των παιδιών που διαρκώ παραβιάζονται, παιδιά που είναι το μέλλον μα και θα δουλεύουν για μα το μέλλον. Αυτά τα παιδιά που βρισκόνται τώρα στο, στην Ευρώπη, είπατε για 6 εκατομμύρια Ρωμά, εγώ νομίζω ότι είναι τουλάχιστον 16 και 100 εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι που δεν είναι Ρωμά. Τουλάχιστον λοιπόν 17 εκατομμύρια είναι παιδιά που ζουν χωρίς ε, επαρκείς συνθήκες ε, υγειονομικής κάλυψης, εκπαίδευσης και όλων των απαραίτητων για μια καλή διαβίωση. Κυρία Σάντους, ευχαριστώ. Εδώ, από ακούσαμε και από τους ομιλητές, μιλάμε για υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ακτιβιστών και ενίσχυση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών. Εδώ ήθελα να μιλήσω λίγο για την κατάσταση στη Μεσόγειο και το πώ ξαφνικά ποινικοποιείται η ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Η διαδικασία κατά τη Ουγγαρία για το μεταναστευτικό, αυτή η δίκη, είναι ένα γεγονός. Όμως δεν είδα η Επιτροπή να αναλαμβάνει δραστηριότερο ρόλο για να καταπολεμήσει αυτά που συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες, να καταδικάσει αυτά που συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες στην ε, ε, Μεσόγειο. Οι νομοθετικές ε, πρωτοβουλίες της Ιταλίας δείχνουν ότι ποινικοποιείται η ανθρωπιστική βοήθεια των με κυβερνητικών οργανώσεων στη φάση της διάσωσης ακόμα και της έρευνας στην πρώτη φάση και μετά της διάσωση των ανθρώπων που ρισκάρουν τη ζωή τους στη Μεσόγειο. Ήθελα λοιπόν να ακούσω από την πλευρά σας τι σκέφτεστε να κάνετε στο, στο διάστημα. Ο κύριος ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ ακριβώ να κάνω την ίδια ερώτηση με τη συνάδελφο Ισαβέλ Σάντο προ την κυρία Μπάρμπαρα Νόλαν, μας είπατε ότι ουσιαστικά έχουν ε, ξεκινήσει διάφορες προσφυγές κατά της Ουγγαρίας και άλλων μελών. Αλλά υπήρξε σαφής παραβίαση του άρθρου 18 του χάρτη ως προς δικαίωμα του ασύλου ε, όταν έκλεισαν τα λιμάνια στην Ιταλία. Μέχρι και σήμερα. Ακόμα κλειστά είναι, είδαμε τις ειδήσει και στην περίπτωση της Μάλτας. Τι δράσεις λοιπόν έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με ε, αυτή τη σαφή παραβίαση του δικαιώματος στο άσυλο. Είναι μια συμπεριφορά που είναι γενικώ αντινομική ε, και αντισυνταγματική κατά των συνθηκών και κατά της εσωτερικής αγοράς. Και σύντομα, ο κύριο Φλάχερτη, αν έχετε να μας πείτε κάτι για την εκπαίδευση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, κυρία Βίσελα, Όχι. Όχι. Thank you, Chair. Director Flaherty, during the... Ε, Βίντσε, ευχαριστώ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, κύριε Φλάχερτη. Είχα δυσκολίες να απαντήσω σε πολίτες που με ρωτούσαν για τα θεμελιώδη δικαιώματα και από αυτόχθονες ε, ε, μειονότητες παρόλο που είναι από, ε, πάνω από 10% του συνολικού πληθυσμού. Ξέρουμε ότι υπάρχει ο θεμελιώδης χάρης, το ξέρουν και εκείνοι, αλλά είναι απογοητευμένοι γιατί δεν εφαρμόζεται στεναρά. Στο μέλλον τι θα γίνει. Και δεύτερη ερώτηση. Ε, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, σχεδιάζει στο προσεχές μέλλον να κάνει μελέτες και συστάσεις σε ό,τι αφορά τις παραδοσιακές μειονότητες. Ε, με τη δεκαετία επέτειο της συνθήκης της Λισαβόνας νομίζω είναι επίκαιρο να γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Η κυρία Πούρεκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις. Όπως γνωρίζουμε όλοι, ε, πριν τεθεί σε ισχύ ο θεμελιώδη χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, πριν από 10 χρόνια, έχει υπογραφεί το λεγόμενο Βρετανικό Πρωτόκολλο με τη Βρετανία και στην Πολωνία, που, ε, λέει ότι δεν εφαρμόζεται σε Βρετανού και Πολωνού πολίτε το σύνολο του χάρτη. Για του Βρετανού ε, ήταν το νομικό σύστημα. Και στην Πολωνία τότε η πρώτη κυβέρνηση της δικαιοσύνης και του νόμου ανησύχησε βαθύτατα για τα αντίπεινα σε Πολωνούς ε, πολίτες. Ε, το έχετε μελετήσει αυτό στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Είδατε όλοι ότι ήρθε ο Επίτροπος Κίνγκ. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας και το εκτιμούμε πολύ. Μερικά λεπτά ακόμα έχουμε. Mrs. please one minute. Κυρία Uh, I'll be speaking in Swedish. Θα μιλήσω σου ειδικά. Ευχαριστούμε για αυτή την πολύ συνολική και διεξοδική παρουσίαση. Αποτελώ ε, μέρος των ανθρώπων που αφορά η παρουσίασή σας, διότι και εγώ είμαι από μια οικογένεια μουσουλμάνων μεταναστών. Ξέρετε ότι υπάρχει διακριτική μεταχείριση κατά των μουσουλμάνων στην Ευρώπη, ιδίω των γυναικών και των παιδιών. Τι γίνεται με αυτέ τι ομάδε του πληθυσμού που συγκεντρώνουν αυτά τα χαρακτηριστικά και σε ποιε περιοχέ. Και μια άλλη ερώτηση. Κάτι το θετικό που αναφέρατε. Πώς μπορούμε να αγωνιστούμε για να εφαρμοστεί οδηγία κατά τη διακριτική μεταχείρισης. Στο επίπεδο του Συμβουλίου υπήρχε μπλοκάρισμα. Πώς μπορούμε λοιπόν να παραμείνουμε σε συμμορφώση με την κάρτα. Ευχαριστώ. Εγώ θα μιλήσω α, ουγγρικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η χάρτα των θεμελιδών δικαιωμάτων προβλέπει συγκεκριμένε αξίε, όπω την ανεξάρτητη λειτουργία του δικαστικού συστήματο, του ίσου μισθού για την ίδια εργασία. Κάποιοι πολιτικοί λένε ότι το σύνολο αυτών των αξιών μπορούν να ερμηνευθούν αλλιώς από κάποιες εθνικές νομοθεσίες και μπορεί να περιοριστούν εφόσον το επιθυμούν κάποιοι. Το θέμα όμως είναι κατά πόσο αυτή η παραβίαση γίνεται συστηματική από, κάποιες, ε, ε, από κάποια δεξιά κόμματα, όπως την Ουγγαρία. I will speak in Polish. Ε, Πολωνικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε που παρουσιάσατε την ε, κατάσταση συνολικά για την εφαρμογή της χάρτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ διρωτώ με το εξής, στο πλαίσιο της μελλοντική μας συζήτησης. Θα μπορεί η χάρτα των θεμελιδών δικαιωμάτων να εφαρμόζεται ώστε να καταπολεμήσουμε το ρατσισμό και την παραπληροφόρηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ του προσκεκλημένου μα για τι παρουσιάσει του. Να σταθώ και εγώ στα δικαιώματα των παιδιών, τα οποία θα είναι πλήρω κάτοχοι θεμελιών δικαιωμάτων, αλλά δεν μπορούν να τα ασκήσουν και να τα προστατεύσουν. Ξέρουμε την φτώχεια των παιδιών, ξέρουμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα βία ε, με του ε, διακινητέ που ασκούν βία κατά των παιδιών των μεταναστών, ε, σωματική βία, η ψυχολογική. Είναι εκτεθειμένα τα παιδιά και υπάρχει και πρόβλημα πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Εκεί έχουμε προβλέψει τις ε, δικονομικές ε, διαδικασίες που πρέπει να προβλέπουν την προστασία των ανηλίκων. Γι' αυτό λοιπόν η ερώτησή μου προς τους προσκεκλημένους μας. Βάσει ποιον όρων ελέγξατε την εφαρμογή της χάρτας σε σχέση με τα δικαιώματα των παιδιών και ε, εάν και υπό ποιε προϋποθέσεις, κυρίως προς τον κύριο Φλάχερτη, μπορείτε να πείτε ότι πραγματικά έχουμε μια σαφή εικόνα για το τι συμβαίνει με τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών. Ευχαριστούμε. Φεστ. Χωρίς μικρόφωνο. Mike, bitte. Jetzt, now. Um, zwei Fragen an Mr. Δύο Διαβάσαμε πρόσφατα σε ένα εβραϊκό έντυπο ότι ε, στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια ε, όσοι Εβραίοι έχουν σκοτωθεί έχουν σκοτωθεί από μουσουλμάνους. Ε, τώρα οι μουσουλμάνοι είναι χειρότεροι εχθή των Εβραίων. Και το δεύτερο που ακούσαμε ω ομάδα που κινδυνεύει είναι οι μετανάστες που πνίγονται στη Μεσόγειο. Τι δουλειά έχει αυτό ε, με ε, τη διάκριση. Αν κάποιος ευρωβουλευτής που έρχεται με το αυτοκίνητό του στις Βρυξέλλες σκοτωθεί σε τροχαίο, τι δουλειά έχει με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τι αξίζει μια τέτοια μελέτη που χειρίζεται τόσο επιπόλαια και τόσο άστοχα τον όρο διάκριση, ο Πρόεδρος. Τώρα, όπως βλέπετε, υπάρχει ένα φάσμα θεμάτων και ερωτήσεων και πραγματικά θα σας παρακαλέσω ό,τι καλύτερο μπορείτε, τρία-τέσσερα λεπτά ο καθένας, όσο το δυνατόν συνοπτικότερα. Διότι ο Επίτροπος Κίνγκ πόσο να περιμένει. Και είναι και πολλά τα σημεία που έχουμε και για τη συνέχεια της ημερήσιας διάταξης. Κυρία Νόλαν, πρώτη εσείς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εντάχει, η ερώτηση για την ψηφιοποίηση. και την τεχνητή νοημοσύνη. Θα έχετε δει ότι η πρόεδρος ε, ακόμα 100 μέρες δεν έχει συμπληρώσει και έχει ήδη προτείνει μια πρωτοβουλία για την τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε συνυπεύθυνοι με την DG Connect για να χτενίσουμε αυτή την νομοθετική πρόταση. Το εξετάζουμε λοιπόν με ιδιαίτερη προσοχή από τη σκοπιά των θεμελιωδών δικαιωμάτων, διότι η τεχνητή νομοσύνη εγείρει σοβαρά θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πρέπει το προ... η πρόταση αυτή νομοθεσία, που θα είναι και κάτι το πρωτοποριακό παγκοσμίω, να γίνει πολύ προσεκτικά. Δεν υπάρχει νόμος που να διευθετεί το θέμα προς στιγμή. Για τι παρατηρήσει τη κυρία Ιντβελτ. Δεν είναι δίκαιο να πούμε ότι δεν εφαρμόζεται τίποτα. Σα διάβασα τι διαδικασίε επί παραβάση, τη λίστα δηλαδή, για, την, ε, για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίω στην Ουγγαρία και την Πολωνία προς στιγμή. Κάτι κάνουμε. Οι υποθέσει βέβαια αυτέ είναι δύσκολε. Χρειάζονται και χρόνο και πάρα πολλή δουλειά και προετοιμασία. Πάντως αυτό που, που κάνουμε, που είναι το καθήκον μας, το κάνουμε. Είμαστε θεματοφύλακε των συνθηκών. Και αναλαμβάνουμε δράση όπου αυτό χρειάζεται. Για το Ταμείο. Είχαμε κάποιες διμερείς ανταλλαγές. Η Επιτροπή προς στιγμήν εφαρμόζει ενεργά όσα απαιτούνται για το Ταμείο. Πιστεύουμε ότι θα χρειαστούμε στην κοινωνία των πολιτών και στην ομάδα των ε, κυβερνητικών οργανώσεων να κάνουμε περισσότερη δουλειά για να ενημερώσουμε. Εκεί επικεντρώνεται το Ταμείο. Εγώ ξέρω ότι θεωρείται ότι πρέπει να πηγαίνουν οι πληρωμές περισσότερο για την ε, διατησία και τη νομική αρρωγή. Οι δικηγόροι Όμω, εφόσον δεν λαμβάνουν και καμία αμοιβή, δεν θα μπορούν και να υποστηρίξουν τι μη κυβερνητικέ οργανώσει για να κάνουν οι ίδιε αυτή τη στρατηγική διατησία, τη δουλειά στρατηγική διατησία που απαιτείται από τι ίδιε. Για την κυρία Γιάροκα. Σα θυμάμαι από ε, τη δουλειά σα στο παρελθόν για του Ρωμά. Για τα δικαιώματα των παιδιών. Ασχολούμαστε με μια συγκεκριμένη ομάδα με τα δικαιώματα των παιδιών. Το συμπεριλάβαμε στη χάρτα. Είναι πολύ σημαντικό τομέα, αλλά είναι μέρο του συνόλου των θεμελιωδών δικαιωμάτων που συμβαίνει με τα παιδιά. Και θα έχετε προσέξει ότι τις επιστολές αρμοδιοτήτων τη ε, ε Πρόεδρου της που επεστάλησαν αυτή την εβδομάδα υπάρχει μια νέα στρατηγική με τα δικαιώματα των παιδιών την οποία θα επεξεργαστούμε σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο για να ενισχυθούν περαιτέρω τα δικαιώματα των παιδιών. ο Μάικλ να απαντήσει στα υπόλοιπα, ε, θα έλεγα. Ευχαριστούμε που είστε σύντομοι. Κύριε Φλάχερτη, ξέρουμε και εσείς πόσο είστε ταγμένος στο σκοπό σας. θα έλεγα τι απαντήσει σα, ε, τι λεπτομερεί, να τι ετοιμάσετε γραπτό και να τις στείλετε με mail, αλλά έχετε και 3-4 λεπτά εφόσον το επιθυμείτε, γιατί έχουμε και τον Επίτροπο Κίν και άλλα σημεία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για την ψηφιοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη. Να διαβεβαιώσω την Επιτροπή ότι είναι πραγματική προτεραιότητα του οργανισμού. Έχουμε επενδύσει στη χαρτογράφηση του θέματο και το τι συμβαίνει με τα δικαιώματα και όσου ασχολούνται με αυτά. Και κάνουμε δύο πράγματα καταρχήν. Πρώτα απ' όλα, χαρτογραφούμε. Βλέπουμε πώ επηρεάζει ήδη η τεχνητή νοημοσύνη τον χώρο των, των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Υπάρχουν πολλά πράγματα που ακούγονται. Το διαδίκτυο, το διαδίκτυο των πραγμάτων, πρέπει να ξεπεράσουμε τους φόβους και τις φήμες που κυκλοφορούν. Επίσης θα χρειαστεί ε, κάποια περισσότερη δουλειά για την αναγνώριση των χαρακτηριστικών ας πούμε ε, και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πριν δύο εβδομάδες ε, είδαμε τι γίνεται με την εφαρμογή της προστασίας των προσωπικών δικαιωμάτων σε συνδυασμό με, με την τεχνητή νοημοσύνη για την ερώτηση της κυρίας τα αφορούσε περισσότερο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από ότι εμένα, την επιβολή του, των όσων προβλέπουν τα νομοθετήματα για τα, για τα θεμελιώδη και τα βασικά δικαιώματα. Ε, αλλά είναι υπεύθυνα τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, δεν βλέπουμε αρκετέ δίκε ή προσφυγέ ε, στι περιπτώσει των ε, εγκλημάτων ή των εκφράσεων μίσου κατά των δημόσιων λειτουργών, α πούμε. Για τα παιδιά θα συμφωνήσω με αυτό που είπε η κυρία Νόλαν. Για τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, η διάσταση των δικαιωμάτων των παιδιών ε, συμπεριλαμβάνεται και εντάσσεται σε όλα όσα κάνουμε. Κοιτάζουμε ιδίω την κατάσταση των παιδιών σε πολύ περίπλοκε περιπτώσει, όπω του μετανάστε. Κυρίω επικεντρωνόμαστε στην κατάσταση των παιδιών όταν κοιτάμε του μετανάστε. Ε, Τι ερχόμενε εβδομάδε, να το πω αυτό στην Επιτροπή σα, θα δημοσιευτεί έκθεση για την επιστροφή ανηλίκων σε τρίτα κράτη. Έχει να κάνει απευθεία με τα δικαιώματα των παιδιών βεβαίω και είναι πολύ σημαντικό σκέλο τη όλη μα δουλειά. Σε ό,τι αφορά τη Μεσόγειο, η κυρία Σάντο το έθεσε, όπω και ο κύριο Φέστ. Είναι θέμα δικαίου, δικαίου τη θάλασσα και του διεθνού ανθρωπιστικού δικαίου. Υποχρεώμεθα και να διασώζουμε ανθρώπους που κινδυνεύουν στη θάλασσα. Και πρέπει να πω ότι πάλι χαρτογραφήσαμε το τι έγινε με τα ε, πλοία που το 2018 δραστηριοποιήθηκαν στη Μεσόγειο και είδαμε ότι ότι καμία απαγόρευση, η απαγόρευση από δεν οδήγησε σε ε, δίκη απαγόρευση του κατάπλου δεν οδήγησε σε δίκη ή νομική προσφυγή. Για τον κύριο Ντεβέσα και την ε, εκπαίδευση των νομικών, να πω ότι δεν υπάρχει πολλή χρόνο. Καλά κάνατε όμω και το θίξατε. Πρέπει να συνεχίσουμε να ε, μορφώνουμε, διότι το ποινικό δίκαιο είναι ένα πράγμα, αλλά είναι και το ανθρωπιστικό δίκαιο πολύ σημαντικό για να αλλάξουμε τι κοινωνίε μα και να μπορέσουμε να εγγράψουμε τι θεμελιώδει αξίε σε όλου του τομεί, καθώ και τα δικαιώματα των παιδιών. Στον κύριο Βίντσε, μιλήσατε για τι εθνοτικέ και γλωσσικέ γλωσσικές μειονότητες. Καλωσορίζω την ερώτησή σα Υπάρχουν. Είναι πραγματικότητα είναι μέρο αυτού του παζλ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, του πολύχρωμου παζλ που έχουμε γύρω μα. Ε, δεν έχουμε ακόμα στα χέρια μα. Αλλά λαμβάνουμε συχνά αιτήματα από εσά για να ολοκληρώσουμε, για να προχωρήσουμε και σε αυτό το χώρο. Και μας ενδιαφέρουν αυτά τα αιτήματα. Πώς βλέπουμε το πολωνικό πρωτόκολλο σε σχέση με τη χάρτα. Δεν το έχουμε αναλύσει ακόμα, πρέπει να σας πω, έτσι απλά, αλλά ευχαριστώ για την ερώτηση, κύριε Αλσαλάμι. Άρχισα να απαντάω στην ερώτησή σα για το πώ κοιτάζουμε το θέμα των παιδιών σε πλαίσιο, στο πλαίσιο των μειονοτήτων, των μεταναστών, αλλά και οι γυναίκε συμπεριλαμβάνουμε αυτά που μας έχουν πει οι γυναίκες, τα διδάγματα από τις εμπειρίες μαζί τους, ειδικά με τις γυναίκες ε, μετανάστηδες, σε όλες τις πολιτικές μας και τις γυναίκες Ρωμά. Ε, εδώ βλέπουμε ότι είναι συνήθως πιο ευάλωτη η θέση των γυναικών και ιδίω σε σύγκριση με τους άντρες. Συμφωνώ για τις οικουμενικές αξίες και όχι απλώς ευρωπαϊκές, είναι οικουμενικές οι αξίες της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και μετά από την, ε, μάλλον από την ε, διακήρυξη την οικουμενική για τα ανθρώπινα δικαιώματα εμπνευστήκαμε και στη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Τώρα, η ελευθερία και η εξάλληψη των εφρέσεων μίσους. Υπάρχουν αυτά. Είναι πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο. Απλώς πρέπει να λάβουμε πολύ πιο σοβαρά υπόψη την εφαρμογή όλων των νόμων και των κανόνων που ήδη διαθέτουμε. Και στον κύριο Φως, Φέστ, για τη χρήση μάλλον για τη συμπεριφορά κατά των μουσουλμάνων. Ε, είδαμε για τη σχέση Εβραίων και Μουσουλμάνων, λοιπόν, εδώ σε κάποιες χώρες δεν είδαμε την, δεν έχουμε δει ακόμα την ειδική αυτή σχέση. Απλώς το τι γίνεται με ομάδες της ακροδεξιάς, εφόσον υπάρχουν ε, συμμετοχές από, μουσουλμανική, από τη μουσουλμανική κοινότητα, αλλά παρά τις μεγάλες μεταναστευτικές μετακινήσεις από το 2015, δεν είδαμε να υπάρχει άμεση σχέση με το ποιοι είναι οι αυτούργοι των εγκλημάτων σε αυτές τις περιπτώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Ε, να πω και εγώ κάτι ως ε, ε συμπέρασμα. Δεν υπάρχει αφιβολία ότι 10 χρόνια μετά από την έναρξη ισχύω ε, του σοβαρού, ε, του, του νομικά δεσμευτικού Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων υπάρχουν βελτιώσεις. Ε, τώρα, οι πραγματικές προκλήσεις είναι το να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο, να ενημερώσουμε για τη σημασία αυτού και το δεσμευτικό χαρακτήρα, νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα αυτού του χάρτη, τόσο για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, όσο και για τα κρατημέλη. Υπάρχει μια αλληλουχία πολύ σημαντικών ε, ε, ε, αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που αποδεικνύουν τη σημασία αυτού του χάρτη ακόμα και υποθέσεις που ξεκίνησαν μετά από μία έφεση νομική καταγγελία η ενέργεια οποιασδήποτε φύσης και να ήταν που ε, υποβλήθηκε και προτάθηκε από, αυτήν, από εδώ, από το Ευρωκοινοβούλιο. Και ε, το Ευρωκοινοβούλιο υπέβαλε στο ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για υποθέσεις όπου ε, η τελική απόφαση αποτελεί πλέον προηγούμενο. Κύριε Λίζε, ε, μια πολύ σύντομη παρατήρηση. Θα σας... Ναι, πολύ σύντομα. Και η κυρία Άντρης και εγώ ε, ε θεωρούμε ότι η κυρία Νόλα δεν απάντησε στις ερωτήσεις ε, που θέσαμε για το τι γίνεται στα λιμάνια. Ίσως μπορεί να μας απαντήσει γραπτός. Αν μπορείτε να δώσετε και τώρα μια σύντομη απάντηση. Αν μας στείλετε επιστολή θα σας ε, απαντήσουμε, αλλά δεν είναι άμεσα ε, δική μου εντολή, δεν εμπίπτει στο δικό μου τομέα, αλλά εάν μας στείλετε επιστολή στην Επιτροπή θα επανέλθουμε από αυτού. Αυτά λοιπόν. Αλλά δεν είναι το τέλος ε, αυτής της υπόθεσης, διότι, όπως είπα, υπάρχουν διάφορα σεμινάρια ε, ε, και ε, συνεδριάσεις που θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα ώστε να ε, εορτάσουμε και να αξιολογήσουμε, να αξιοποιήσουμε αυτόν τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ όλους και θα προχωρήσουμε καλωσορίζοντας τον Επίτροπο King για το δεύτερο σημείο. Συνεχίζουμε, μην χαλαρώνετε. Ευχαριστούμε, Επίτροπε Κίνγκ, ε, που ήρθατε. Ε, είναι θέμα ασφάλειας αυτό και ο Επίτροπος Ασφάλειας προφανώς, ο κύριος ε, Κίνγκ, αρμόδιος για την Ένωση Ασφάλειας. Έχουμε υπόψη μας ότι η πολιτική ασφαλεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατοχυρώνει μια σειρά από εργαλεία για να ενισχύσουμε την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών τα έχουμε συζητήσει αυτά τα θέματα και πάρα πολύ για την παραπληροφόρηση και την κυβερνοασφάλεια ε, στις επικοινωνίες και ακριβώς για αυτό το θέμα θα μας μιλήσει σήμερα ο Επίτροπος Κίνγκ. Εμείς συζητήσαμε την επιρροή ε, της παραπληροφόρησης στις εκλογικές διαδικασίες και στην ίδια τη δημοκρατία τελικά. Τώρα όμως βλέπουμε νέες τεχνολογίες, όπως είναι τα deep fake, η τεχνητή νοημοσύνη, οι πλατφόρμες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ε, οργιάζει η παραπληροφόρηση και απειλεί τη δημοκρατία σε όλα τα κράτη-μέλη. Έχουμε συζητήσει για πρακτικές, βέλτιστες πρακτικές, κανόνες δεοντολογίας και συμπεριφοράς, αλλά και αυτά αποδείχτηκαν ανεπαρκή. Θα μας παρουσιάσει λοιπόν ο Επίτροπος Κίνγκ τα μελλοντικά βήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τη μελλοντική νομοθεσία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στο κυβερνοχώρο και τα δίκτυα 5G ε, που είναι τώρα έτσι, η τελευταία λέξη της μόδας ε, στις νέες τεχνολογίες και ενδεχομένως επηρεάζουν την επιβολή ε, του νόμου και την πρόσβαση των διοκτικών αρχών σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Θα σας δώσουμε το λόγο κύριε Επίτροπε και μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση. Πρώτα οι συντονιστές παρακαλώ σύντομα και οι δυνατόν ε, και τα υπόλοιπα μέλη. Γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και είναι και αρμοδιότητά μας. Καλώς ορίσατε Επίτροπε. Ευχαριστώ που με δέχεστε και πάλι. Α, πριν ακριβώς ε, τις καλοκαιρινές διακοπές αρχίσαμε να συζητούμε για κάποια από τα θέματα και τις, επι, τις ε, επιπτώσεις ε, των νέων τεχνολογιών, τις νέες συμπεριφορές επίσης που καταχρώνται αυτής της τεχνολογίας και με χαρά είδα ότι προτείνατε τη σημερινή συζήτηση. Βεβαίω, είναι μια ελαφρώς ιδιαίτερη περίοδο αυτή τη στιγμή, περίοδος αυτή τη στιγμή γιατί γίνονται πολλά, γίνονται πολλές συζητήσεις για τη νέα Επιτροπή αλλά υπάρχουν και πολλά που θα πρέπει να κάνουμε από τώρα μέχρι τα τέλη του Οκτωβρίου και γι' αυτό μαζί θέλω να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε όλα αυτά τα θέματα. Η πρόεδρος μελλοντική της Επιτροπής έχει πει ότι η ψηφιοποίηση μεταμορφώνει τις αγορές μας και τον τρόπο ζωής μας και ότι θα πρέπει να ε, το εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε περισσότερο μέσω των ε, big data και των διαφόρων άλλων ε, ευκαιριών ενώ ταυτόχρονα, εφόσον θέλουμε να αποκομίσουμε τα ωφέλη, θα πρέπει να ασφαλιστούμε ενάντια στους ενδεχόμενους κίνδυνους. Δηλαδή, να βρούμε δηλαδή πώς θα μειώσουμε τους κινδύνους που προέρχονται όταν κάποιοι προσπαθούν να παρέμβουν στην τεχνολογία μας ή να την καταχραστούν για να μας βλάψουν. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να σκεφτούμε όχι μόνο την οικονομική και βιομηχανική πτυχή όλων αυτών, όπου είναι όντως πολύ σημαντική, αλλά και την πτυχή, τη διάσταση της ασφάλειας, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες μας και ολόκληρες μας τις κοινωνίες από τους κακόβουλους φορείς από ευρωπαϊκή άποψη. Αυτό σημαίνει ότι ε, πρέπει να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε τις σωστές επιλογές Άρα λοιπόν θα πρέπει να ε, μεριμνήσουμε ώστε, θα πρέπει, ε, ώστε η νέα τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί με καλόβουλο τρόπο και να μην μπορούν οι κακόβουλοι φορείς, όπως είπαμε, οι παίχτες να μπορούν να το εκμεταλλευτούν. Να αρχίσω με το 5G. Το ανέφερε ε, η πρόεδρος εδώ. Ε, είναι πάρα πολύ κρίσιμο για να προστατεύσει από επιθέσεις, από κατασκοπία, από αναγκαστική μεταφορά τεχνολογίας ε, και είναι και πολύ σημαντικό όσον αφορά την γεωπολιτική κατάσταση. Για να το καταφέρουμε αυτό θα πρέπει να ενεργήσουμε από κοινού σε ολόκληρη την Ευρώπη για να εντοπίσουμε και να καλύψουμε αδυναμίες ε, που μπορεί να υποβαθμίσουν την συλλογική μας ασφάλεια. Γι' αυτό και νωρίτερα φέτος η Κομισιόν έκανε μια σύσταση που ξέθεσε μια προσέγγιση για να αναπτυχθεί το δίκτυο 5G με προηγούμενες γενναίες ε, τηλεπικοινωνιών 2, 3 και 4G η τιμή και το κόστος ήταν τα βασικά μας μελήματα ενώ για το 5G θέλουμε ως πρώτο μέλημα να βάλουμε την ασφάλεια όσον αφορά την λήψη αποφάσεων. Η, η ανάγκη για ε, συλλογική δράση είναι προφανής εφόσον ε, μιλάμε για ευρωπαϊκή δομή και γι' αυτό και έχουμε φτιάξει μια τριφασική προσέγγιση, σε τρεις φάσεις δηλαδή. Ε, πρώτον, εντοπισμός κινδύνων, αυτό έχει ήδη ολοκληρωθεί και όλα τα κρατημέλη υπέβαλαν ε, τις ε, αναφορές τους. Δεύτερη φάση είναι που εξέλιξε τώρα και πρέπει να συνδυάσουμε δηλαδή αυτές τις ανησυχίες και να σχηματίσουμε ευρωπαϊκή εικόνα για τους κινδύνους και να αρχίσουμε να διατυπώνουμε στρατηγικές για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, πράγμα που θα κάνουμε μέχρι το τέλος του έτους. Προχωράμε λοιπόν καλά. Η επόμενη τυπική, το επόμενο τυπικά στάδιο θα είναι τον, στα μέσα Οκτωβρίου που εγώ και η Μαρία Γκαμπριέλ θα ε, αναφέρουμε τι αποκομίσαμε από το διάλογο με τα κράτη-μέλη για τους κινδύνους και προσβλέπουμε σε κάποια από τα μέτρα που θα προταθούν για να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους. Ε, τώρα, εσείς ως ε, ενεργά μέλη της πολιτικής συζήτησης στη χώρα σας, ε, είσαστε και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ποιοι είναι οι δυνητικοί κίνδυνοι της παραπληροφόρησης και πώς μπορεί να, η παραπληροφόρηση να παρασύρει ολόκληρες δημοκρατικές διαδικασίες, εκλογές, να διχάσει κοινότητες στις κοινωνίες μας. Για να προσπαθήσουμε να αποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις, η Κομισιόν έχει αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες. Έχουμε εκδώσει ανακοινωθέν για την ε, αντιμετώπιση της επιγραμμικής παραπληροφόρησης το 18, τον περασμένο Σεπτέμβριο ένα πράγμα δράσης και ένα μια δέσμη ε, πακέτο, ένα πακέτο δηλαδή μέτρων το πέρυσι θα πρέπει οι ιδιωτικοί και οι δημόσιοι να αναλάβουν δράση, η το εθνικό επίπεδο, οι επιγραμμικέ πλατφόρμες, οι διαφημιστές, οι δημοσιογράφοι, τα, οι όμιλοι ενημέρωση οι ε, καθηγητές, δάσκαλοι, όλοι πρέπει να συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια. Ζούμε στην ψηφιακή εποχή τελικά όταν ε, κανείς το σκεφτεί δεν έγινε και τόσο θεαματική παραπληροφόρηση στη διάρκεια των ευρωεκλογών. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξε παραπληροφόρηση. Όχι. Πολύ παραπληροφόρησε μάλιστα και κυκλοφόρησε. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, Υπήρξαν ε, έκθεσεις, ε, εκθέσεις, αναφορές ότι στη Γερμανία η επιγραμμική πρόθεση ενός συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος αντιπροσώπευε 86% ε, όλων όλης της κομματικής δραστηριότητα στο Facebook προς τη, τη διάρκεια της εκλογικής εκστρατείας. Τέσσερις φορές περισσότερα σχόλια, έξι φορές περισσότερο το μερίδιο όλων των άλλων κομμάτων Πολλά από αυτά τα like και τα μοιρασιά προέρχεται από ύποπτους λογαριασμούς με δύο αρχικά συνήθως που είναι συνήθως στην τύχη και ο ένας ε, λογαριασμός ε, έκανε like στον άλλον και τούμπαλ είναι για να και, το, και, και το έκαναν share για να διαδοθεί περισσότερο και Πάει λέγοντα. Άρα λοιπόν έτσι γίνεται μια μεγάλη κλίμακα προπα... Ε, προπαγάνδα παραπληροφόρηση. Εάν λοιπόν ε, είναι ύποπτα αυτά τα, ε, αυτοί οι λογαριασμοί με δύο τυχαία και κεφαλαία γράμματα, έχουμε πρόβλημα. Εγώ δεν θέλω να το δεχτώ αυτό ως βάση για την πολιτική μας ζωή στην Ευρώπη. Γι' αυτό και ε, ήρθαμε σε επαφή με τις μεγάλες πλατφόρμες ώστε να υπογράψουν ε, τον κώδικα για την παραπληροφόρηση που οροξητικοποιήθηκε πέρυσι το Σεπτέμβριο. Έχουμε ε, Mozilla, Facebook, Twitter, καθώς και το διαφημιστικό τομέα και τους εκπροσώπους, όλοι δεσμεύτηκαν να τα κάνουν αυτά. Έκτοτε και η Microsoft μπήκε και υπέγραψε αυτόν τον κώδικα διοντολογίας. Υπάρχουν διάφορες δεσμεύσεις, σε 15 τον αριθμό και παρακολουθούμε τι συμβαίνει και ελέγχουμε ε, τακτικά οποτεδήποτε γίνονται εκλογές. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τι γίνεται. Στα μέσα Σεπτεμβρίου περιμένουμε οι ίδιοι οι, οι συνυπογράφοντες στον κώδικα να υποβάλουν αναφορές ε, σχετικές προς την Επιτροπή. Έχουμε ε, επίσης ανεξάρτητα τρίτα μέρη ε, συμβούλους που θα μας αναφέρουν επίσης, θα κάνουν επίσης εκθέσεις αναφοράς για το τι συμβαίνει. Με βάση όλα αυτά η Κομισιόν θα ανακοινώσει μια πρώτη ε, αναφορά για το πώς προχωράει η εφαρμογή αυτού του κώδικα πριν τα τέλη Οκτωβρίου. Τελευταίο στάδιο θα είναι η πλήρη αξιολόγηση υπό τη μορφή ανακοινοθέντου τη Κομισιόν που αναμένεται να εκδοθεί στι αρχέ του επόμενου έτου με περαιτέρω ε, διαβουλεύσεις με τους ειδικού του ίντερνετ και τα κράτη-μέλη. Όπως έχω πει και προηγουμένως, η Επίτροπος ε, Γκαμπριέλ είπε ότι αν όλα αυτά δεν είναι ικανοποιητικά, πιστεύουμε ότι θα πρέπει η Κομισιόν να να προτείνει περαιτέρω ενέργειες. Τώρα, για την χειραγώγηση της παρα, παραπληροφόρησης επιγραμμικά, το Google, το Twitter και το Facebook έχουν προβεί σε δράση και αυτό το καλωσορίζουμε και μοιράζονται περισσότερα στοιχεία καθώς και τη δημιουργία ε, προέβησαν στη λειτουργία πολιτικών κατευθυντηρίων γραμμών. Ε, θα πρέπει οι πλατφόρμες να δίνουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες ε, ώστε να επιτρέπεται η ταυτοποίηση των επιγραμμικών ε, ε, παιχτών και ποιον στοχεύουν, να δημοσιεύουν τα στοιχεία από τα κρατημέλη και να δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες να καταλάβουν πιο εύκολα ποιοι είναι αυτοί οι φορείς και πώς μπορούμε να έχουμε πρόσβαση, βέβαια σύμμορφα με τους κανόνες της προστασίας των δεδομένων για να γνωρίζουμε καλύτερα τι συμβαίνει. Υπάρχουν διάφορες νομοθετικές και άλλου είδους προτάσεις που έχουν υποβληθεί στα κράτη-μέλη, μας, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό το έχουν εξετάσει με ένα έγγραφο περί επιγραμμικών βλαβών. Στη Γαλλία έχουν πιέσει ώστε οι πάροχοι του ίντερνετ να είναι πιο υπόλογοι και Επίσης, στους μήνες πριν τις εκλογές, ε, φέραμε τις εκλογικές επιτροπές και τους ειδικού ε, κυβερνοασφάλειας σε ένα ενισχυμένο δίκτυο, ε, σε επαφή δηλαδή μέσω ενός ενισχυμένου δικτύου, ώστε να μοιραστούν τις πρακτικές και να οικοδομήσουν περισσότερη ανθεκτικότητα και αντίσταση η σημασία της διαφάνειας είναι πολύ μεγάλη, ιδιαίτερα στην ε, πολιτική διαφήμιση. Θα επανέλθουμε λοιπόν με μια έκθεση προς εσάς για τις εκλογές, πώς πήγαν αυτές αργότερα μέσα στο φθινόπωρο. Επίσης, νωρίς φέτος ε, δημιουργήσαμε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Ένωση ώστε να μπορούμε να εντοπίζουμε και να, ε, τις ε, εξατήσεις παραπληροφόρησης όσο γίνεται πιο έγκαιρα. Στη διάρκεια αυτών των εκλογών δεν είδαμε να γίνεται κάποια μεγάλη εξατία παραπληροφόρησης, όμως και εμείς είχαμε αυξημένες επαφές και συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά και να δημιουργήσουμε και ένα κόμβο για έρευνα και ανάλυση σε συνεργασία με διεθνούς εταίρους μαζί με τον ΝΑΤΟ και τους G7. Τα τελευταία δύο χρόνια κινητοποιήσαμε μια κοινότητα ελεγκτών ε, στοιχείων, ε, ερευνητών που βοηθούν στην ανάλυση εκστατιών παραπληροφόρησης και που προσπαθούν να σχεδιάσουν απαντήσεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή αντιμετώπιση. Κάνοντας έτσι, έχουμε φτιάξει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την παραπληροφόρηση μέσω της, του προγράμματος Connecting Europe. Ε, και για να γίνει αυτό θα πρέπει και οι πλατφόρμες των κοινωνικών μέσων να κάνουν τη δική τους δουλειά, να παρέχουν δηλαδή ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα για αυτούς τους έμπιστους ελεγκτές στοιχείων, ώστε να μπορούν και αυτοί να κάνουν την έρευνά τους και να δίνουν καλύτερες απαντήσεις και αντιμετώπιση, ενώ βεβαίω ε, θα εξασφαλίζουμε την τήρηση των επαγγελματικών και ηθικών προδιαγραφών. Χρειαζόμαστε και εργαλεία για να χειριστούμε αυτέ τι πληροφορίε. Μέσω του Horizon 2020 έχουμε επενδύσει πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ με την Κομισιόν ώστε να ε, ε, μπορέσουμε να χειραγωγήσουμε τι νέε τεχνολογίε και να επιταχύνουμε την ανάπτυξη διαφόρων project και εταιρικών σχέσεων, καθώ και τη δημιουργία επαφών ανάμεσα στου ερευνητέ, ε, επιχειρηματική κοινότητα και ε, τις πλατφόρμες. 16 ε, δις προτείνουμε δε για το επόμενο PDP, ώστε να στηριχθούν τέτοιου είδους μέτρα και άλλα μέτρα που προωθούν το ποιοτική δημοσιογραφία, την ελευθεροτυπία και τον πλουραλισμό. Έχουμε προχωρήσει, έχουμε σημειώσει πρόοδο, έχουμε ακόμα καλά, πολλά να κάνουμε. Ε, με ευτυχής που είναι στην ατζέντα τα θέματα αυτά και στο νέο επίτροπο ε, και της ε, ε, μελλοντικής Προέδρου έχουμε, έχει ας πούμε προβλέψει μια ευρωπαϊκή συντονισμένη προσέγγιση για τα ανθρώπινα και ε, την ανθρώπινε επιπτώσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και βεβαίως όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά ώστε να έχουμε ένα ασφαλές ψηφιακό μέλλον για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Επίτροπε Κίνγκ. Μεταξύ των υβριδικών απειλών αναφερθήκατε στις επενδύσεις και τη δουλειά που έχει κάνει για να θεωρητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν άνθρωποι που επενδύουν εκατομμύρια στην παραπληροφόρηση και θα πρέπει και είναι απαραίτητο να μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις για αυτό το θέμα που είναι τόσο λεπτό ε, στο πλαίσιο των υβριδικών απειλών για τις δημοκρατίες μας. Θα κάνουμε ένα πρώτο γύρο ερωτήσεων με τους συντονιστές ή τους εκπροσώπους τους και αν δεν απατώμε θα μιλήσει πρώτος ο κύριος Λέναρς από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και Επίτροπε Κίνγκ επικεντρωθώ στο 5G. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Κανείς δεν αρνείται τις ενδεχόμενες χρήσεις και τη χρησιμότητα, αλλά υπάρχουν και θέματα ασφαλείας. Και έχει δύο όψεις αυτό. Την ασφάλεια του δικτύου που αναφέρατε ε, λεπτομερώς, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την Huawei, ε, την εταιρεία την κινέζικη, τις κινέζικες μυστικές υπηρεσίες κτλ. Την περασμένη φορά τέσσερι χώρε νομίζω έχασαν την προθεσμία για τι μελέτε αντικτύπου, τώρα από ό,τι άκουσα όλε τα έκαναν. Δεν είναι φυσικά ευρωπαϊκό θέμα, είναι παγκόσμιο το 5G. Πώ έχει λοιπόν η συνεργασία εκεί τη Ευρωπαϊκή Ένωση με συναδέλφου, ας πούμε από την Αυστραλία, τις Ηνωμένε Πολιτείε, Διότι τι ίδιε ανησυχίε συμμερίζονται και αυτοί και η κατάσταση είναι η ίδια. Ε, δεύτερον, δεν έχει να κάνει μόνο αυτό με την ασφάλεια του ίδιου του δικτύου, αλλά τι κάνουν οι υπηρεσίες ασφαλείας, οι αρχές και πώς μπορούν να λειτουργούν στην εποχή του 5G. Θυμάμαι το έγγραφο θέσεων της Ευρωπόλ τον Απρίλιο, που έλεγε ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνονται νόμιμες παρακολουθήσεις τηλεφώνων. Ε, το, ε, το IMS, ας πούμε, ε, τώρα γίνεται παροχημένο ε, για ανθρώπους που αλλάζουν συνέχεια κάρτες SIM και τα λοιπά, για την κρυπτογράφηση. Ε, όλα τα στοιχεία, τα νέα του 5G δυσκολεύουν πάρα πολύ τις διοκτικές αρχές να κάνουν τη δουλειά τους με νόμιμο τρόπο, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή. Ερωτώ λοιπόν, τι μπορούμε εμείς να κάνουμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι προτίθεται να κάνει, για να βεβαιωθούμε, επειδή τρέχουν οι εξελίξεις, είναι ραγδαίες, να είναι έτοιμε οι διοκτικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν έρθει η τεχνολογία αυτή να εργαστεί σε ένα πεδίο και περιβάλλον 5G και να μας διατηρεί ασφαλή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Η συντονίστρια των ε, σοσιαλιστών, η κυρία Ζίπελ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα αρχίσω κι εγώ από το 5G. Εκπλήσω με λίγο, διότι τον τελευταίο μήνα άκουσα από διάφορες χώρες ότι «Α, σπουδαίο, τέλεια, έρχεται το 5G, ε, πιο γρήγορο ίντερνετ για όλους» και τώρα ακόμα ότι υπάρχουν και προβλήματα που δεν είναι μόνο το 5G, αλλά και η κρυπτογράφηση. Και εδώ έχουμε πρόβλημα, γιατί η κρυπτογράφηση είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο για τον οικονομικό κλάδο και για τις εταιρείε, αλλά για τους δικηγόρους, δημοσιογράφους, καταγγέλλοντες, μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Δεν μπορούμε να απορρίπτουμε την ιδέα της κρυπτογράφησης. Σε ποιο βαθμό όμως χρειάζεται για την επιβολή του νόμου και για τις διοκτικές αρχές υπάρχουν άλλες λύσεις, υπάρχει άλλος τρόπος να ενημερώνεται η αστυνομία. Και ε, θέλω να το συνδέσω αυτό με ένα άλλο ερώτημα. Όλο και περισσότερο συζητούμε για τις νέες τεχνολογίες και τίνουμε να λέμε ε, να συνεργαστούμε με ιδιωτικές εταιρείες που έχουν την τεχνογνωσία. Από την άλλη, ακούω από κρατικές αρχές, ε, δικαιοσύνη και αστυνομία, ότι δεν έχουν τους εμπειρογνώμονες που χρειάζονται ε, της πληροφορικής. Ε, ε, άρα αυτό θέτει ένα ερώτημα. Όταν συνεργαζόμαστε με ιδιώτες, έχουμε εμεί τον έλεγχο των όσων κάνουν εκείνοι, όταν οργανώνουν εκείνοι τις τεχνολογικές εφαρμογές για μας. Γίνονται τέτοιες συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βρούμε έναν τρόπο να αυξήσουμε τις τεχνικές, τεχνολογικές γνώσεις, τις δικές μας διοκτικές αρχές και κρατικές αρχές. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Από την ομάδα Renew Europe. Ε, ε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you, um, for, uh, Renew Europe. Uh- Ευχαριστώ από το Renew Europe Ευχαριστώ, Επίτροπε Κίν. Καταλαβαίνω ότι έχουμε τεράστια προβλήματα με την ε, ε, χειραγώγηση των ψηφοφόρων και την παραπληροφόρησή τους. Πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο και με το δημοψήφισμα του 2016 το είδαμε αυτό. Είχαμε και αποδεικτικά στοιχεία ότι υπήρξαν τεράστιες εκστρατείες παραπληροφόρησης και στο διαδίκτυο και από blog και αν έχουμε γενικέ εκλογέ στο Ηνωμένο Βασίλειο και πλέον δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι θα πρέπει να γίνει. Από τα μέτρα πρόληψη που αναφέρατε, πολλά ε, έρχονται πολύ αργά να κάνουν κάτι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι μπορεί να κάνει για να βοηθήσει τις εθνικές ε, εκλογικές επιτροπές να προβλέψουν ένδικα μέσα όταν υπάρχει σαφής ε, απόδειξη, όταν υπάρχουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία ότι υπάρχει οργανωμένη προσπάθεια απάτης και η κυβέρνηση δεν λαμβάνει δράση κατά της εκλογικής απάτης ή της νοθείας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Στρίκ. Από τους Πρασίνους, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τον Επίτροπο Κίνγκ για τη διεξοδική παρουσίαση. Από την πλευρά των Πρασίνων να τονίσω ότι και εμείς υποστηρίζουμε εφόσον αναγνωρίζουμε την ανάγκη να προστατεύσουμε τους πολίτες από την παραπληροφόρηση και τις εκφράσεις μίσους. Αλλά υπάρχει και η ανάγκη, απ' την άλλη, να προστατεύσουμε την ελευθερία της έκφρασης και την πρόσβαση στην ε, πληροφορία την ίδια. Στην Επιτροπή, λοιπόν, πώς μπορείτε να εξισορροπήσετε τις δύο αυτές αντίρροπες δυνάμεις. Τι μέσα θα εκδιπλώσετε για να πετύχουμε αυτή την εξισορρόπηση και όσο, σε ό,τι αφορά την διαφάνεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πιέσει για τη διάσταση της διαφάνειας σε πολιτικές διαφημίσεις λόγου χάρη. Όμως εδώ χρειάζονται κανόνες απτοί για να υπάρξει και διαφάνεια. Τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι απτές ε, και συγκεκριμένες προτάσεις θα κάνει για την επιβολή του νόμου σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ταρντίνο από την ομάδα ID. Ευχαριστώ. Διότι ήδη ανέγνωσα την παρέμβασή μου σε προηγούμενη φάση. Οπότε τώρα θα είμαι κάπως συνοπτικότερη. Απευθείας μια ερώτηση. Το είπαν και οι συνάδελφοι. Σε ό,τι αφορά την παραπληροφόρηση, η Επιτροπή μας είπε τι έχει γίνει ως τώρα, ιδίως με εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Και σε συνεργασία με ιδιωτικού φορεί. Βλέπω όμω τα περισσότερα κράτη-μέλη, τα μέτρα, να μην είναι, τα μέτρα να μην είναι επαρκή για να καταπολεμήσουμε τι ψευδεί ειδήσει και την παραπληροφόρηση. Όπω είπαν λοιπόν και οι συνάδελφοι. Τι μέτρα θα λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για το άμεσο χρονικό διάστημα μπροστά μα. Υπάρχουν κράτη-μέλη που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα σε περιόδους προεκλογικής εκστατείας αλλά και μετά ε, στην παραπληροφόρηση, στη διάδοση ψευδών ειδήσεων. Πώς θα αναχαιτήσουμε αυτό το φαινόμενο ενδεχομένως και με πρόβλεψη νομοθετικών μέτρων. Ευχαριστώ πολύ. Από την ομάδα ECR, ο κύριος Προκατσίνη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Επίτροπο. Για την παραπληροφόρηση μια ερώτηση η πολιτική, εμπορική πληροφόρηση και επικοινωνία ε, λαμβάνει πλέον χώρα, το γνωρίζουμε όλοι, στο διαδίκτυο σε μεγάλο βαθμό. Τα τελευταία όμως χρόνια, με αυτά που έχουμε δει να συμβαίνουν, δεν θεωρείται ότι μόνον μία δημόσια αρχή με αστυνομικές, θα έλεγα, αρμοδιότητες ή έστω δικαστικές νομικού χαρακτήρα μπορεί να διαγράφει ή να εξαλείφει ιστότοπους ή λογαριασμούς χρηστών από τα κοινωνικά δίκτυα. Είναι στα χέρια των ιδιωτικών εταιριών όλα αυτά που βρίσκονται και εκτός ευρωπαϊκών συνόρων δεν θεωρείτε ότι θα, υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει μια δημόσια αρχή, κρατική αρχή που να έχει μεγαλύτερη αρμοδιότητα σε αυτό το τομέα. Και για το 5G. Δεν κατάλαβα πολύ καλά την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το πρόβλημα με τη highway. Εδώ ε, ο αντιπρόεδρος της εταιρεία που είναι υπεύθυνο για την περιοχή της Ευρώπης γιόρταζε και με λίγο προκλητικό τρόπο απέναντι έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών την έναρξη της περιπέτειας της Huawei στην Ευρώπη. Η δική σα θέση λοιπόν από αυτού ποια είναι. Ευχαριστώ πολύ. Η, η κυρία Πελτιέ, αν δεν απατώμε. Παρακαλώ. Πρέπει να σας πω ότι θα κλείσει ο κατάλογος των ομιλητών για το δεύτερο γύρο όταν τελειώσουν οι συντονιστές γιατί έχουν ζητήσει πάρα πολλοί συνάδελφοι το λόγο και θα σας διαβάσω τον κατάλογο. Αν υπάρχει κανένα πρόβλημα. El señor Peter, el señor Estrugaru, el señor Tudorache, el señor Ross, el señor Chebowski, la señora Kinichi, el señor Fest, el señor Breyer, Κλείνει ο κατάλογος, αν δεν έχω κάνει κανένα λάθος. προχωρά... Ε, είναι για το δεύτερο γύρο των ομιλητών. Κύριε Απελτή, έχετε το λόγο. Με ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Θα ήθελα απλώς να σε ευχαριστήσω ε, την προσοχή να σε πιστήσω την προσοχή σε μια κατάσταση που διαρκεί στα κράτη-μέλη και στην Ευρώπη και ποιες είναι οι προτάσεις σας θέλω να μάθω σχετικά με το άρθρο 13 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Μιλάτε για τα παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση στο σχολείο. Εγώ σκέφτομαι τα παιδιά των μεταναστών, τα παιδιά με αναπηρία. Ε, είναι θεμελιώδης δικαίωμα και στη ΛΥΜΠΕ θα πρέπει να ασχοληθείτε εσείς με αυτό το θέμα που είναι πραγματικά θεμελιώδες. Ευχαριστώ. Δέκα λεπτά τώρα έχει ο κύριος Κίνγκ για να απαντήσει στους συντονιστές. Παρακαλώ. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά μετά με τις ερωτήσεις μπορεί να καλύψω κάποια πράγματα στο δεύτερο γύρο. Αν κάτι ξεχάσω, φροντίστε να το συμπληρώσετε στι επερωτήσει. Για το 5G πρώτα απ' όλα. Έχετε δίκιο. Για την ασφάλεια του συστήματος υπάρχουν κάποια θέματα. Τεχνικά ζητήματα και το πώς συμπεριφέρεται το δίκτυο, το σύστημα, πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς. Για τα της ασφαλείας. Το μελετούμε το θέμα, θα ολοκληρωθεί ανάλυση μέχρι το τέλος του χρόνου, σε συνεργασία με όλα τα κράτη-μέλη. Και αυτά είναι ζητήματα που βρίσκονται βεβαίω στην καρδιά του ζητήματο τη εθνική ασφάλεια. Οπότε όλα τα κρατη έχουν ε, κάθε λόγο να, συνεργα... να ενώσουν τι δυνάμει του και να συνεργαστούμε. Θα δημοσιοποιήσουμε όλα τα πορίσματα του κάθε βήματος και στην ε, επικοινωνιακή μας πολιτική. Έχουμε και εξωευρωπαϊκούς εταίρους, είπα Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, συνομιλούμε με όλους για να αντλήσουμε εμπειρίες και διδάγματα. Έχουμε, για να απαντήσω και στον κύριο Προκατσίνη, έχουμε ευθύς εξ αρχής καθορίσει ότι θέλουμε να ακολουθήσουμε κάποιες αρχές που έχουμε ορίσει εκ των προτέρων. Δεν θέλουμε όμω να πούμε ότι αναγκαστικά θα καταλήξουμε σε αρνητικά αποτελέσματα. Θα δούμε τι αποδεικτικά στοιχεία μπορούμε να συλλέξουμε και πώ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Αλλά αυτή εξ αρχή έχουμε καθορίσει το ότι θέλουμε στο τέλο τη όλη προσπάθεια να καταλήξουμε σε συλλογική συμφωνία με τα κράτη-μέλη για προϊόντα, υπηρεσίε ή παρο... που μπορούν να παράσχουν ασφάλεια και να μπορούμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους. Δεν μας νοιάζει ποιος θα είναι αυτός ο πάροχος ή ποια υπηρεσία, αλλά αν κάτι δεν είναι ασφαλές στο τέλος της όλης εξέτασης, θα το πούμε ανοιχτά, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να λάβουν μέτρα, να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Αυτό ισχύει για οποιαδήποτε εταιρεία, και τη Highway και οποιονδήποτε άλλο. Τώρα, για διαφορετικές συμπεριφορές ε, στο όλο αυτό σύστημα και δίκτυο και το πώς τα πράγματα μπορεί κάπως να σκοτεινιάσουν λόγω της κρυπτογράφησης ή των τεχνικών διαδικασιών για τις νέες μορφές επικοινωνίας που θα δημιουργηθούν. Τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Έχει βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησής μας αυτό με τα κράτη-μέλη και με τους ειδικευμένους οργανισμούς όπως η Europol. Πρέπει να μιλήσουμε και με τις αρχές επιβολής του νόμου και να δούμε πώς ακριβώς θα υπάρχει σωστή εφαρμογή των κανόνων. Δεν μπορούμε να ζούμε σε ένα σκοτεινό κόσμο, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε και τη σημασία της κρυπτογράφησης στις ζωές μας. Ούτως ή άλλως. Προστατεύει η κρυπτογράφηση τι ζωέ μα. Δεν θα ήθελα να ζω σε ένα κόσμο χωρί κρυπτογράφηση ό,τι αφορά με τα τραπεζικά μου Πρέπει να βρούμε λοιπόν έναν τρόπο να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την εγκεκριμένη, την ελεγχόμενη πρόσβαση για τις αρχές επιβολής του νόμου ας πούμε, χωρίς όμως να υπονομεύουμε την ακαιρεότητα των συστημάτων κρυπτογράφησης που εμείς οι ίδιοι έχουμε δημιουργήσει, αλλά να μην ανοίξουμε παραθυράκια για παράνομη πρόσβαση σε εγκληματίες ή παραβάτες. Αυτή είναι η πρόκληση. Η πρόκληση είναι ξεκάθαρη και η δυσκολία που έχουμε. Δεν είναι πολύ δύσκολο να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Δύο πράγματα λοιπόν πρέπει να πω προ στιγμή. Έχουμε κάνει δύο πράγματα στην πράξη. Πρώτα απ' όλα για την υποστήριξη των αρχών επιβολή του νόμου, συμπεριλαμβανομένη τη ε, Europol, να δούμε πώ οι ίδιοι μπορούν να αναπτύξουν τι τεχνικέ του γνώσει και δυνατότητε και συνεργαζόμαστε και με τη διεθνή κοινότητα. για το τι είδου πρότυπα και προδιαγραφέ μπορούμε να καταρτήσουμε για τη χρήση του 5G και άλλων τεχνολογικών μέσων. Θέλουμε ουσιαστικά να φροντίσουμε οι αρχέ επιβολή του νόμου να μην βρεθούν στην απέξω, αποκλεισμένοι από την όλη αυτή διαδικασία. Φροντίζουμε λοιπόν να προσφέρουμε κι άλλα κονδύλια στη Europol για να κοιτάξει πώ θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτά σε συγκεκριμένε συσκευέ, τα λάπτοπ, στα κινητά τηλέφωνα. Έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων ε, με συμμετέχοντε από τι αρχέ επιβολή των κρατών μελών που μπορούν να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίε, με δύο εργαλειοθήκε που θα μπορούν να χρησιμοποιούν νομίμω. Έχουμε δύο ερευνητικά προγράμματα για να δούμε τρόπου αντιμετώπιση των θεμάτων τη νόμιμης και εγκεκριμένης κρυπτογράφησης, της αντιμετώπισης της παράνομης, χωρίς να διακυβευθεί η κανονική κρυπτογράφηση και προωθούμε και νομοθεσία για την ταχύτερη και ε, ευκολότερη πρόσβαση των δικαστικών και νομοθετικών των δικαστικών και ε, αρχών, των διοκτικών αρχών στις στα αποδεικτικά στοιχεία. Για την παραπληροφόρηση. Όπως είπατε αρκετοί από εσάς, Πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία διαγραφής παράνομου περιεχομένου, εκφράσεων μίσους και προσπαθειών παραπληροφόρησης, διατηρώντας ταυτόχρονα τις αρχές που προσπιζόμαστε, ξεκινώντας από την ελευθερία της έκφρασης. Εμείς το θεωρούμε εφικτό. Και το τελευταίο 1,5 χρόνο αυτό που ξεκινήσαμε να κάνουμε και ελπίζουμε να το συνεχίσει και η επόμενη Επιτροπή είναι να διακρίνουμε μεταξύ παρανόμου περιεχομένου, δηλαδή προνογραφικό περιεχόμενο που εκμεταλλεύεται τα παιδιά, εκφράσεις μίσους, τρομοκρατικό περιεχόμενο. Να διακρίνουμε λοιπόν μεταξύ παρανόμου περιεχομένου. Δεν είναι ελεύθερη από τις έκφρασεις αυτό, είναι παράνομο. Ξεκάθαρη γραμμή διαχωρισμού. Με άλλα πράγματα Υπάρχει ένα φάσμα μορφών επικοινωνίας, εκφράσεων μίσους, που δεν μπορούμε να τα επιβάλλουμε νομοθετικά, αλλά με συμφωνίες κυρίων κάποιοι προτείνουν νομοθετικά μέτρα και σε αυτό το τομέα και μετά υπάρχει και η διάσταση της παραπληροφόρησης της ηθελημένης διάδοσης και διασποράς ε, ψευδών πληροφοριών και ειδήσεων στο διαδικτυακό χώρο. Εδώ πρέπει να προωθήσουμε την διαφάνεια. Υπάρχει μια σειρά από μέτρα που προβλέψαμε στον κώδικα, σχεδιασμένα για να προωθήσουν τη διαφάνεια, ώστε να δούμε πώς τι γίνεται με τους ψεύτικους ε, λογαριασμούς, τα bot και τους ε, ε, πώς μπορεί ένας ελεγκτής να τα παρακολουθεί και να τα επιθεωρεί. Έχουμε κάνει σε εθελούσια βάση όμως κάποια πρόοδο, αλλά όπως είπα και το πρωί δεν είναι αρκετή αυτή η πρόοδος ακόμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει τι έχει γίνει σε σχέση με το παρελθόν. Και αργότερα μες στη χρονιά όταν κάνουμε την επισκόπησή μας θα πούμε ότι η πρόοδος δεν είναι ακόμα αρκετή. Ενδεχομένως να χρειαστούν και περαιτέρω μέτρα νομοθετικά, δεσμευτικά, που να επικεντρώνονται τους κανόνες για τη διαφάνεια. Δεν θέλουμε κανόνες για το τι είναι καλό ή κακό περιεχόμενο, τι είναι νόμιμο ή ένομο, ε, παράνομο. Σε περιπτώσεις ε, πολιτικής ή προεκλογικής επικοινωνία, πρέπει να ξέρουμε ε, να διασφαλίσουμε την διαφάνεια για τις πηγές. Οι πολίτε να ξέρουν αυτό που βλέπουν, από πού προέρχεται, πού προέκυψε Υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη μεμονωμένα μέσω του δικτύου που σα παρουσίασα. Για το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί υπήρξαν και συγκεκριμένα για την Αγγλία. Έχουμε έναν πολύ δραστήριο συνεργάτη στην υπηρεσία για την διαφάνεια των πληροφοριών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει ε, ασχοληθεί πολύ σοβαρά με τις έρευνες για τα περιστατικά που αναφέρατε. και σε συνεργασία με άλλου φορεί πληροφοριών και δικτύων ε, σε εθνικό επίπεδο. Για την ερώτηση και πάλι του κυρίου Προκατσίνη για τι δημόσιε αρχέ που θα μπορούσαν να αναλάβουν δράση εκείνε αντί για τι ιδιωτικέ εταιρείε. Έχουμε συνεργασία με ιδιωτικέ εταιρείε, διότι αυτή είναι και η φύση του αντικειμένου. Δυστυχώ είναι ιδιωτικό ο τομέα που πρέπει να καλύψουμε. Σε εθελοντική βάση υπάρχει αυτή τη στιγμή η συνεργασία μας και δεν θα πρέπει βεβαίω να αποφύγουμε να προβλέψουμε και νομοθετικού κανόνε όποτε πρέπει. Παράνομο τρομοκρατικό περιεχόμενο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει και ελπίζω να συμφωνήσουν και οι, όλοι, οι υπόλοιποι συνομιλητέ μα στου τριμερεί διαλόγου ότι όντω πρέπει να υπάρξουν νέοι κανόνε. Οι δικαστικέ αρχέ, οι αρχέ επιβολή του νόμου θα πρέπει να μπορούν να παρέμβουν όταν εντοπίσουν ότι υπάρχει σαφώ παράνομο τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο και οι ιδιωτικές εταιρείες θα, θα είναι υποχρεωμένε να δώσουν κάποια απάντηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Επίτροπε Κίνγκ. Και τώρα θα προσπαθήσουμε συνήθω να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μιλήσετε όλοι. 15 τουλάχιστον έχετε ζητήσει το λόγο. Μισή ώρα έχουμε προβλέψει στην ημερήσια διάταξη για το υπόλοιπο αυτού του θέματος. Φτάνει Λοιπόν, ένα λεπτό καθένας για να προλάβουμε να ακούσουμε όλους. Ετοιμαστείτε να πυροβολήσετε μέσα σε ένα λεπτό, να εκτοξεύσετε την ερώτησή σας. Έλκα. Ο κύριος Κρίς ε, Πέτερς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, short the was already... Ε, θα είμαι πολύ σύντομος, γιατί έχει γίνει ήδη ερώτηση για το 5G και την ασφάλεια. Ξέρω ότι ζητήσατε από όλα τα κράτη-μέλη να στείλουν ε, τα εθνικά τους ε, σχέδια για την εκτίμηση κινδύνου και τον Οκτώβριο θα βγάλει την ανακοίνωση. Ανησυχώ λίγο πρέπει να πω για το τι θα πρέπει να αναλυφθεί ως πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αυτό το θέμα. First, in Belgium, for example, we are... Στο Βέλγιο πρώτα απ' όλα ε, είμαστε τώρα στην τελική φάση να το κάνουμε πολύ χειροπιαστό το 5G. Και στη συνέχεια, αν δούμε ε, τις εκτιμήσεις κινδύνου, τις εθνικές που σας έχουν στείλει όλα τα κράτη-μέλη, θα υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία από χώρα σε χώρα. Ερωτώ λοιπόν, το ξέρω ότι δουλεύετε πολύ γρήγορα, αλλά θα προλάβετε, θα υπάρξει κάποια ε, πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε η ασφάλεια να είναι πολύ στενή και πολύ γρήγορα να έρθουν όλα αυτά. Κύριο Κλοντ Μωράη, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Επίτροπε για όλη αυτή τη δουλειά που κάνετε. Πραγματικά συζητούμε την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και το 5G σε ένα εθελοντικό πλαίσιο για την αδειοδότηση. Και συζητήσαμε και με τον επικεφαλής της ΕΝΗΣΑ στην Επιτροπή ε, Βιομηχανίας για τα παγκόσμια στάνταρτ, αλλά όλη η Επιτροπή Ιτρε μιλάει ε, και η βιομηχανία για ε, υποχρεωτική πιστοποίηση. Ξέρετε, είμαι αναπληρωτή στην Επιτροπή Ήτρε και παρακολούθησα τις συζητήσεις. Για να μην πολυλογώ, δεν είναι καλύτερα να ε, χρειαστεί υποχρεωτική αδειοδότηση πιστοποίηση παρά να περιμένετε μέχρι το 2023 για την παραπληροφόρηση. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι νέοι βουλευτές ότι εσείς έχετε κάνει πάρα πολλά για θέματα επιγραμμικά και μη ε, που έχουν να κάνουν με ε, τη διαφάνεια, με διάφορους λογαριασμού κτλ. Και ρωτώ, κερδίζουμε σε αυτή τη μάχη και στο Ενωμένο Βασίλειο και αλλού. Έχουμε εξωτερικές παρεμβάσεις σε εκλογές. Δεν χρειάζεται να πω σε λεπτομέρειες. Τι να κάνω σε ένα λεπτό κερδίζουμε αυτή τη μάχη. ή Πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Στην Ολομέλεια την άλλη εβδομάδα θα το συζητήσουμε. Τι θα πούμε για την επέμβαση εκλογές. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα σας ρωτούσα και για τον Brexit, αλλά σηκώθηκε σφυρί. Ε, αν θέλετε... Thank you, Mrs. Thank you, Chair. Να το δούμε διμερώσα. Ε. Η κυρία Στρουγκάριου. Ε, μιλήσατε για το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Δεκεμβρίου του 2018. Ε, και μια πολύ συγκεκριμένη σειρά ερωτήσεων. Μπορείτε να μας δώσετε παραδείγματα για το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ε, για το 2019, για τις πρόσφατες εκλογές. Αναφερθήκατε σε μια κοινότητα ελεγκτών δεδομένων, fact-checkers. Πόσους έχετε δηλαδή και πόσους θα έχετε στο μέλλον. Και τρίτον, priorities and three ε, ποιες είναι οι τρεις προτεραιότητές σας και ε, πρώτη γραμμή για την Μελλοντική Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπράιερ. Uh, Δύο ερωτήσεις για το 5G και την ασφάλεια. Γνωρίζουμε ότι τμήματα του δικτύου θα ανήκουν σε κινέζικες εταιρείες και ξέρουμε ότι οι hacker έχουν χακάρει ε, παγκόσμια δίκτυα για να παρακολουθούν ε, μερικούς ε, συγκεκριμένους ανθρώπους. Εσείς πώς σκοπεύετε να ενισχύσετε. Θέλετε να είναι ενισχυμένο και με κρυπτογράφηση το δίκτυο ή θέλετε να μπορείτε να κάνετε υποκλοπές και παγιδεύσεις, γιατί και τα δύο δεν γίνονται. Ε, στη συνέχεια ακούμε διάφορες προτάσεις από διάφορες γενικές διευθύνσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μία από τη δική σας γενική διεύθυνση λέει ότι σκέφτεστε Ε, ε, μήπως ε, κλείνετε λογαριασμούς όταν έχουμε ρητορική μίσους ή κακόβουλη. Μέχρι τώρα είχατε άλλη τακτική. Τώρα σκέφτεστε να του κλείνετε του λογαριασμού. Ο κύριο Φέστ. Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμη κύριε Επίτροπε Κίνγκ. Φοβάμαι λίγο όταν ακούω τι ομιλίε σα. Λέτε, υποτίθεται ότι στη Γερμανία υπήρξε διαδικασία παραπληροφόρηση και μιλάτε για ύποπτου λογαριασμού Facebook δεν έχετε αποδείξεις ότι είναι αυτόματα bots, αλλιώς θα μιλούσατε για bots και όχι για ύποπτους ε, λογαριασμούς. Εκεί όμως που δεν έχετε αποδείξεις ισχυρίζεστε ότι ήταν ε, κακόβουλοι ε, από κάπου. Αν το γράφατε αυτό σε εφημερίδα θα σας απέλυαν γιατί ανακατεύετε σχόλια με γεγονότα και απόψεις το κράτος δικαιώνει σε καλά χέρια στα χέρια σας. Μάλλον το αντίθετο φαίνεται από αυτά που μας λέτε και οι προτάσεις σας για το ε, fact-checked που είναι και συγκαλυμμένη ε, λογοκρισία. Αυτά έρχεται να επιβεβαιώσουν όσα εγώ ε, πιστεύω. Ευχαριστώ. Να, ευχ... να συγχαρώ τη Μεγάλη Βρετανία να έχει κόσμο και ανθρώπους σαν και εσάς μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στο μέλλον τους. Είναι πολύ θλιβερή ημέρα σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι η τελευταία φορά που θα σας εδώ ως Επίτροπος, αλλά ελπίζω ο διάδοχός σας να είναι εξίσου επάξιος, ε, ε, μάλλον ε, καλό στα καθήκοντά του, γιατί αν ήταν η τελευταία σα παρουσίαση ω Βρετανό Επιτρόπου, ήταν, θα μπορούσε η Μεγάλη Βρετανία να είναι περήφανη για σα. Είστε φοβερό εμπειρογνώμων, πάρα πολύ καλό ρήτορα και φοβερό ε, γνώστη του αντικειμένου. Πραγματικά ελπίζω να βρεθεί κάποιο αντάξιό σα. Έχουμε ακούσει όλη αυτή την ε, καυτή κουβέντα για την ε, κινέζικη εταιρεία, τη Highway, και για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες την κατασκοπία των πολιτών της Ευρώπης ενδεχομένως. Αυτό θα ήθελα να σχολιάσετε. Ευχαριστούμε. Μας θυμήσατε σε όλους το γνωστό ποίημα του Μαρκ Τουέιν. Τα νέα και οι ειδήσει για το θάνατό μου μου φαίνονται κάπως πρόημα, λέει. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω και πάλι ογκρικά. Τα τελευταία χρόνια στην Ουγγαρία είχαμε πάνω από 100 ιστοτόπους που φαίνεται να είχαν διασυνδέσεις με ρωσικές πηγές και διευθύνσεις. Ρωσικά IP. Αυτή η ιστοτοπία, αυτές οι σελίδες είχαν τέτοιο περιεχόμενο που ε, ουσιαστικά ε, στρέφονταν κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη να την αποδυναμώσουν. Στην Ουγγαρία υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα όμως. Αυτές οι ιστοσελίδες Ε, χρησιμοποιούνται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και διωγγώνεται η παρουσία τους ε, γιατί εξυπηρετούν την ε, κυβερνητική πολιτική και τα κυβερνητικά ελεγχόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι υπάρχει μια προσπάθεια αποσταθεροποίησης. Τι μπορεί να κάνει γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί έχει να πει. you, um, Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ Επίτροπε για την παρέμβασή σας. Ε, λέει ο κ. Στοντόρα, θα μείνω και εγώ στο 5G και έρχομαι στις ερωτήσεις αμέσως γιατί πολλοί συνάδελφοι με κάλυψαν. Ε, σε ό,τι αφορά ε, τη δεύτερη και την τρίτη φάση της τριφασικής που μας ε, παρουσιάσατε και ιδιαίτερα την τρίτη φάση, ποια εργαλεία σκέφτεστε να προτείνετε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να βασίζονται στην κοινή εκτίμηση κινδύνου που θα κάνουν τα κράτη-μέλη στη δεύτερη φάση. Πόσο ισχυρά πιστεύετε ότι θα είναι αυτά τα εργαλεία, τι θα είναι συστάσεις, προδιαγραφές ή μήπως θα βάλετε και ε, κάποιες απαιτήσει για τους διαγωνισμούς ε, που θα κάνουν τα κράτη-μέλη. Γιατί τίνω να πιστεύω ότι ορισμένα κράτη-μέλη έχουν προχωρήσει, έχουν προκηρύξει ήδη τους διαγωνισμούς και έχουν αναθέσει και μερίδια της αγοράς σε αυτές τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογίες και άλλα κράτη-μέλη τώρα είναι στο στάδιο της προκήρυξης των διαγωνισμών. Εσείς λοιπόν θα τους βάλετε κάποιες απαιτήσει γιατί έχει σημασία αυτό. Και ε, τελευταίο, ε, μεταξύ αυτών των απαιτήσεων θα είναι η διακυβέρνηση για τις εταιρείες που ε, θα υπάρχουν κάποιοι ιδεοντολογικοί κανόνες και διαφάνεια. Θα μιλήσω λαδικά, λέει ο κ. Ο στόχος που περιγράφει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να δημιουργήσει ένα ανοιχτό πεδίο τύπου ε, χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, χωρίς. Ε, αλλά υπάρχει πρόβλημα εδώ. Εσείς μιλάτε για ανεξαρτησία και ελευθερία, αλλά θέλετε να το κάνετε αναμειγνιόμενοι στο πεδίο το μεντιακό. Ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα, υπάρχουν και πόροι για τρένα δημοσιογράφων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα Πώς θα το χειριστεί, πώς θα εξασφαλίσετε ε, την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης και την ανεξαρτησία των ίδιων των ελεκτών, των fact-checkers. Κύριε Σπιλτσίκ. Uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, το ακούσατε επανειλημμένο στις ερωτήσεις μας. Δεν θεωρούμε ότι έχουμε κάνει αρκετή πρόοδο. Μπορείτε να εντοπίσετε έναν τομέα που θεωρείτε το πλέον προβληματικό. θα ήταν καλό για, το, για τη διαδοχή του Οκτωβρίου και επειδή μπορεί να μην σας ξαναδούμε εδώ ε, για να γνωρίζουμε τι θα κάνουμε και στις ακροάσεις. Επίσης, έχουμε 28 κράτη-μέλη με διαφορετικές πολιτικές ό,τι αφορά την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Βλέπετε και διαφορετική κατανομή των κονδυλίων και των πόρων μεταξύ των κρατών μελών ενδεχομένω. Μήπω αυτέ οι αποκλήσει είναι ένα πρόβλημα, μήπω χρειάζεται διαφορετική διαίρεση των πόρων για να ενισχύσουμε τα κράτη-μέλη που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη να αντιμετωπίσουν την παραπληροφόρηση. Ευχαριστούμε κυρία Κινίτσι. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ και τον Επίτροπο Κίνγκ που μα ε, έδωσε τόσο σοβαρέ πληροφορίε για τι πρωτοβουλίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τη ασφάλεια και την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών μέσων, ιδίω του 5G και όλο ιδιαίτερω με τι ανησυχίε που έχει γύρει η δυσκολία αστυνομικών και δικαστικών ερευνών, τις οποίες ανέφερε η Europol. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τον Επίτροπο Κίνγκ. Επειδή μα είπατε ότι έχετε και συνομιλίε με τι Αμερικανικέ Αρχέ, μπορείτε να μα πείτε κάτι παραπάνω για τα μέτρα που ενδεχομένω θα μπορούσε να εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίω στη διάσταση τη πρόληψη και για να αντιμετωπίσει την ενδεχόμενη χρήση του 5G από πλευρά ε, εγκληματικών και τρομοκρατικών οργανώσεων. Τι μα έχει διδάξει, μάλλον όπω μα έχει διδάξει ως τώρα η πείρα, ε, η εμπειρία μα, ε, είναι ήδη πολύ πιο μπροστά από εμά συνήθω στη χρήση των τεχνολογικών μέσων. Ευχαριστούμε και τώρα κυρία Αντάμοβιτς. Θα μιλήσω πολωνικά. Η παραπληροφόρηση και οι ψευδεί ειδήσει. Σε σχέση με το διαδίκτυο, πολλέ φορέ χρησιμοποιούνται σε μια προσπάθεια αποσταθεροποίησης και προκειμένου να δημιουργήσουν ε, ε, ε, εσωτερικέ διαμάχε που έχουν προκληθεί έξωθεν και σε περίοδο προεκλογικών εξτρατείων ιδίω. Είναι ένα επικίνδυνο όπλο. Ο προσελητισμό, ο φανατισμό τη κοινωνία και η χειραγώγηση των πολιτών. Πώ μπορούμε λοιπόν να προστατεύσουμε τα δημοκρατικά καθεστώτα. Η ερώτησή μου είναι πώ μπορούμε αυτό το επικίνδυνο όπλο να το αναχαιτήσουμε. Τι μπορούμε εμεί να κάνουμε βλέποντας ότι κάποιες φορές τα εθνικά δίκαια σε αυτόν τον τομέα δεν είναι αρκετά για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Επίσης, για τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται θα μπορούσε να προβλεφθεί κάποιο είδους διαδικασία για την κατάργηση αυτών των πλατφορμών εφόσον έχουν παράνομο περιεχόμενο. Εγώ, ακαδημαϊκός και ερευνήτρια, ξέρω ότι υπάρχουν πολλέ τέτοιε περιπτώσει και θα πρέπει να προστατεύουμε σε κάθε περίπτωση την ελευθερία τη έκφραση Επίτροπε, ξέρετε ότι ε, κάναμε επιτάχυνση για να προλάβουμε, διότι ε, το σημείο αυτό προβλεπόταν στις 11 ε, και 4 και αμέσως μετά έχουμε κοινή συνεδρίαση με τα μέλη της Επιτροπής των Δικαιωμάτων των Γυναικών και της Ισότητας των Φίλων. Συμβαίνει συστηματικά αυτό. Έχουμε συνεργασία με την Επιτροπή ΦΑΜ, ως Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, Οπότε θα μιλήσουμε και με τον αρμόδιο επίτροπο για τα θέματα καταπολέμησης διακίνησης ανθρώπων. Ε, μας μένουν 13 λεπτά. Ε, είναι αρκετό χρόνο. Προσπαθήστε να απαντήσετε στο φάσμα των ερωτήσεων που σα έχουν τεθεί. Το λόγο, Επίτροπε Ευχαριστώ. Ίσως τα τελευταία μου 13 λεπτά. Ελπίζω πως όχι. Λοιπόν, έγινε άλλη μια ερώτηση για τη Huawei. Και πάλι, εμείς δεν ξεκινάμε με προκαταλήψεις. Θα κάνουμε τη δουλειά που πρέπει, θα κάνουμε την ανάλυση που πρέπει και αν ανακαλύψουμε ότι υπάρχουν ε, κίνδυνοι, ε, είναι πολύ δύσκολο να σκεφτούμε πώς θα τους διαχειριστούμε ή πώς θα τους αντιμετωπίσουμε. Για συγκεκριμένες υπηρεσίες ή συγκεκριμένους ε, προμηθευτές θα το πούμε. Δεν είμαι σε θέση τώρα να πω ότι θα είναι συγκεκριμένη η τάδε πηγή κινδύνου ή όχι. Όταν θα φτάσουμε στο τέλος αυτού του έτους, για τη συζήτηση για το τι προτείνουμε να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα χρειάζεται να είμαστε σε θέση να εξηγήσουμε και να αιτιολογήσουμε τις προτάσεις μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εάν δηλαδή θέλουμε να μας στηρίξει ο κόσμος και να διαχειριστούμε και όχι να κρυφτούμε για το γεγονό ότι μάλλον θα χρειαστεί να χειριστούμε μια δύσκολη συζήτηση με κάποιου από του διεθνεί μα εταίρου. και συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τη ΣΥΠΑ αλλά μπορεί να έχουμε διαφορετική προσέγγιση ε, σε αυτό. Να έχουμε, έχουμε μια δύσκολη και περίπλοκη ε, σε σχέση με την Κίνα. Είναι δύσκολο να εξηγήσουμε και να αιτιολογήσουμε τα συμπεράσματα στα οποία φτάσαμε στο τέλος του έτους. Και αυτά τα συμπεράσματα θα στηριχτούν από τα κράτη-μέλη. Αυτά θα αποτελέσουν μια... Θα ξεκινήσουν μάλλον με μια σειρά προτινόμενων μέτρων που θα μπορούσαν να ληφθούν ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε και να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους. Είναι αυτό το δυναμικό μας πλαίσιο για τη λήψη των μέτρων, το οποίο ήδη υπάρχει το έχουμε ε, αναφέρει στην αρχική σύσταση ότι το υπάρχον νομικό κείμενο που επιτρέπει τα κρατημέλη να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους για το 5G και να λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια. Δεν χρειάζεται νέα νομοθεσία, χρειάζεται συζήτηση για το κατά πόσο πρέπει να, λεφθούν, να προβλεφθούν νέα μέτρα. Αλλά δεν τα χρειαζόμαστε για να καλύψουμε το θέμα της ασφάλειας. Τα μέτρα τα οποία τώρα εξετάζονται σε ορισμένα κράτη-μέλη και τα οποία γι' αυτόν τον λόγο δεν θα με εντυπωσίαζε αν κάποιες από αυτές τις ιδέες αναφέρονταν στις προτάσεις μας για πράγματα που μπορούν να γίνουν από κοινού σε και την Ευρώπη περιλαμβάνουν την ενίσχυση των, των εφαρμογών ώστε οι φορείς τηλεπικοινωνιών να εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία των δικτύων τους, προηγούμενα καθεστώτα προηγούμενη έγκριση για την ανάπτυξη συγκεκριμένου εξοπλισμού ή απαιτήσει ελέγχου, δοκιμών μάλλον, ε, ή υποχρεώσεις ελέγχου συγκεκριμένων τμήματων των ε, δικτύων, απέτηση ελέγχων ε, για τους παρόχους εξοπλισμού, αλλά και τους εξωτερικούς συνεργάτες. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε από κοινού και δημόσια θα εξηγήσουμε γιατί τελικά κρατάμε μία την άλλη θέση. Υπάρχει και μία διάσταση πιστοποίησης σε όλα αυτά και αυτό ε, ε, ε, το εξηγώ και στον κύριο Μωράης. Όπως γνωρίζετε, είναι υπό εξέλιξη συζήτηση που στον νέο οργανισμό κυβερνοασφάλειας όσον αφορά τα δίκτυα πιστοποίησης, το 5G είναι ένας από τους τομείς όπου χρειάζεται να προχωρήσουμε και αυτή η εργασία έχει ε, δικό του ε, χρονικό περιθώριο για το 5G. Δεν πρέπει να καθυστερήσουμε, πρέπει να μπορέσουμε αυτό το δίκτυο να το ε, χρησιμοποιήσουμε με βάση τα όσα ήδη σας περιέγραψα. Τώρα, τα σχόλια που κάνω είναι βασισμένα σε στοιχεία. Δεν θέλω να κάνω πίσω σε όλα αυτά. Δεν είναι το μόνο παράδειγμα που μπορείτε να βρείτε. Το ανέφερα ένα παράδειγμα στη Γερμανία και ε, νομίζω πως ανέφερα και άλλα παραδείγματα την τελευταία φορά που συζήτησα μαζί σας και από άλλα κρατημέλη. Το να προσπαθούμε να είμαστε διαφανείς για αυτά τα παραδείγματα είναι νομίζω πολύ σημαντικό. Είναι το πρώτο βήμα για να κατανοήσουμε το πρόβλημα και να ε, το αντιμετωπίσουμε. Ε, θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε πίσω από τα παραδείγματα αυτά ή να μην τα αναδείξουμε. Υπάρχουν διότι είναι εξωτερικοί φορείς που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την παραπληροφόρηση. Ας πούμε, έγινε μια ερώτηση για τις ρωσικές, ε, ρωσικούς σύνδεσμους. Έχουμε μια ε, ομάδα που παρακολουθεί τις εξαιτίες παραπληροφόρησης υπέρ του Κρεμλίνου. Μπορείτε να φαντάζεστε ότι είναι παλιό αυτό το πρόβλημα, αλλά αυτή η ομάδα μόλις, μόλις εξέδωσε για φέτος τον όγκο της οργανωμένης παραπληροφόρησης υπέρ του Κρεμλίνου, που ήταν διπλάσιος από πέρσι. Ε, δεν μειούνται λοιπόν το πρόβλημα, αλλά άλλοι, και άλλοι φορείς μπορεί να έχουν μάθει από αυτό τη ρωσική, το ρωσικό βιβλίο, ε, εγχειρίδιο. Οπότε πρέπει να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε όλα είναι και περισσότερη ανθεκτικότητα απέναντι στην παραπληροφόρηση από όπου και άμα αυτή προέρχεται. Ο κ. Μωράης αναφέρθηκε επίσης ε, και ε, στην πρόκληση των ε, ψευδών λογαριασμών. Υπάρχουν δύο τομείς όπου δεν έχει συμβεί πρόοδος μέχρι στιγμής. Ο πρώτος είναι θα πρέπει να είναι ακριβώς το θέμα των ψευδών ε, λογαριασμών και των bots. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Το Facebook δημοσίευσε τεράστια νούμερα για τον αριθμό των ψευδών λογαριασμών που κατέβασαν αλλά επίσης οι ίδιοι δημοσίευσαν ότι ο αριθμός των ψευδών λογαριασμών στο δική τους πλατφόρμα ε, συνεχίζει να αυξάνεται. Οπότε ο καθαρός αριθμός ψευδών λογαριασμών παρά όλες τις προσπάθειες είναι περίπου 124 εκατομμύρια που εκείνοι έχουν εντοπίσει στην πλατφόρμα τους. Μου φαίνεται τεράστιο νούμερο. Αν δούμε τώρα τη δραστηριότητα bot σε άλλες, σε άλλες πλατφόρμες, πάλι οι δείκτες είναι ότι ο όγκος της δραστηριότητας board, δηλαδή ρομπότικη δραστηριότητα, ε, και επίσης αυξάνεται. Και εκεί πρέπει να δράσουμε. Αλλού που πρέπει να σημειωθεί πρόοδος, και εδώ αυτό συσχετίζεται με τους ελεγκτές στοιχείων που σας είπα, είναι το πόσο ανοιχτές είναι οι πλατφόρμες ε, στην στον ανεξάρτητο έλεγχο. Και πάλι το Facebook ε, έχει κάνει καλή δουλειά γιατί έχει βελτιώσει τις πληροφορίες που προσφέρει για το πώς αντιλαμβάνεται το τι γίνεται στις πλατφόρμες του. Αλλά διάφοροι ανεξάρτητοι ερευνητές είπαν ότι βρίσκουν πιο δύσκολο να έχουν πρόσβαση εκτός του Facebook σε στοιχεία που παλιότερα μπορούσαν να αναλύσουν. Αυτό δεν είναι σωστό. Καλωσορίζω το πρώτο βεβαίως, αλλά θα ήθελα να υπάρξει πρόοδος και στο δεύτερο. Δηλαδή, οι πλατφόρμες να ανοίξουν περισσότερο στον ανεξάρτητο έλεγχο. Δεν είναι αποδεκτό οι ίδιοι να βαθμολογούν ε, πώς τα πήγαν, ε, να βαθμολογούν τον εαυτό τους. Επίσης με ρωτήσατε σοβαρές και λεπτομερείς ερωτήσεις για το σύστημα έγκυρης προειδοποίησης και το δίκτυο των ελεγκτών στοιχείων. Σύντομα, δεν έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης ε, στις εκλογές, αλλά ήταν ένα σύστημα για γρήγορη ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ε, όμως το επόμενο στάδιο είναι να ε, μπορέσουμε να αναπτύξουμε ανθρώπινους πόρους, ε, ε, διανοητικούς πόρους, να συνεχίσουμε να οικοδομούμε και να μοιραζόμαστε τις γνώσεις και να οικοδομήσουμε και τη διεθνή συνεργασία στο ΝΑΤΟ και στο G7. Τώρα, οι ελεγκτέ των στοιχείων. Οι ελεγκτέ των στοιχείων με του οποίου συνεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι 38 οργανώσει σε 17 κρατημέλη. Συμμετέχουν και άλλοι, αλλά εκεί είναι. αυτό είναι ο πυρήνα. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι αυτοί οι ομάδες έχουν πάρει ένα μέρος που θα, θα, θα ασκούσαν ε, λογοκρισία είναι απόλυτα διαφανής για, στη δουλειά που κάνουν και στην κατανόηση που έχουν των όσων γίνεται. Θέλουμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε αυτήν την κοινότητα των ελεγκτών των στοιχείων και γι' αυτό όπως ανέφερα θα χρηματοδοτήσουμε από την, το πρόγραμμα Διευκόλυνση για την Ευρώπη μια νέα Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Παραπληροφόρηση που θα, στόχο θα έχει να βοηθήσει τον κόσμο που εργάζεται για αυτά τα θέματα, τους ανεξάρτητους ελεκτές στοιχείων και ε, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να μπορούν να μοιράζονται ε, τις πληροφορίες που συλλέγουν. Χρειάζεται να έχουμε οι πλατφόρμες να ασχοληθούν και αυτές με αυτή την εργασία, αυτού του είδους τη δουλειά. Οι ερευνητές θα πρέπει να είναι σε θέση με τις πλατφόρμες ε, να ε, δημιουργούν κάποιο ρύθμιση για ε, ασφαλή πρόσβαση στα στοιχεία που έχουν οι πλατφόρμες για την παραπληροφόρηση ώστε να κατανοούν το φαινόμενο καλύτερα. Αυτό είναι μια πρόκληση και είναι πρόκληση για τώρα αλλά και για την επόμενη Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε για τη συντομία και για την προσπάθεια να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, σε μία-μία. Είναι προφανές ότι εδώ τώρα δεν σας αποχαιρετούμε, δεν σας κάνουμε τον επικίδιο ε, του Επιτρόπου. Σας είπα ηρωνικά προηγουμένως αυτό που είπε ο Μαρκ Τουέιν. Είστε ολοζώντανος, δεν έχετε παραδώσει το πνεύμα. Ε, ε ίσα ίσα ε, έχετε μακρά παράδοση τέτοιων επιδόσεων ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε αυτή την πολιτική ασφαλείας. Ο κύριος Δεχόφσκι, ο συνάδελφός μας, είχε δίκιο πάντως όταν μας θύμισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να είναι υπερήφανο που σας έχει ως επίτροπο αρμόδιο για αυτά τα θέματα όλα αυτά τα χρόνια. Really You have a, Πραγματικά, ε, είστε διπλωμάτης καριέρας, ε, και μεταξύ αυτών δεν δείχνετε και πολύ τα συναισθήματά σας ε, όταν ε, μιλάτε δημόσια, αλλά όλοι είμαστε εκλεγμένοι πολιτικοί και μπορούμε να δείξουμε κάποια συγκίνηση τη στιγμή που σας φύγουμε το χέρι και σας λέμε ευχαριστούμε Επίτροπε εκεί. Θα τα ξαναπούμε λέει ο Επίτροπος. Ελπίζω. Λοιπόν, είμαστε ακριβώς στην ώρα μας για το επόμενο θέμα στην ημερησία που σας είπα. Ε, ε, υποδεχόμαστε και μέλη της Επιτροπής των Γυναικών και Ισότητας των Φίλων, δικαιωμάτων των γυναικών καλύτερα, και Ισότητας των Φίλων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα περιμένουμε λίγα λεπτά να βρουν τις θέσει του και να καθίσουν. Σα ευχαριστώ για την υπομονή σα. Well, as we said, we move on. Λοιπόν, όπως είπαμε, προχωρούμε. Couple of points to go through. Έχουμε ακόμα κάποια θεματάκια να δούμε στη σημερινή συνεδρίαση. Καλωσορίσατε λοιπόν εσείς τα μέλη της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φίλων, ΦΑΜ, μαζί με τα εναπομείναντα μέλη τα δικά μας. Καθίστε παρακαλώ. Και ετοιμαστείτε. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Είναι κοινή η συζήτηση όπως σας είπα Rights and Gender Equality, namely Είναι τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και της Επιτροπής ΦΑΜ για να συζητήσουμε την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, δεύτερη έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται στις ενέργειες για την καταπολέμηση εμπορίας ανθρώπων του 2018 όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 20 της Οδηγίας 2011 κάθετος 36 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της. Έχουμε και πάλι την τιμή ε, να υποδεχόμαστε εδώ στο Προεδρείο την κυρία Μαρία Βασιλιάδου, όχι για πρώτη φορά, τη γνωρίζουμε όλοι μας. Είναι συντονίστρια κατά του τράφικινγκ της εμπορίας ε, ανθρώπων και έρχεται να μας παρουσιάσει τη δεύτερη έκθεση. Επίσης έχουμε μέλη της Επιτροπής ΦΑΜ, όπως είπα επανειλημμένα προηγουμένως, έχουμε την Αντιπρόεδρο Οχένια Ροντρίγκες Παλόπ. Δεν ξέρω αν θα θέλετε να πείτε δύο λόγια πριν πάρει το λόγο η κυρία Βασιλιάδου. Παρακαλώ. Θέλετε. Okay. Ε, yes, yes. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Επιτροπή Γυναικών εδώ και καιρό τονίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι θύματα της εμπορίας, δυσανάλογα. Ε, και αυτό είναι βία, διαρθρωτική βία, διαρθρωμένη κατά των γυναικών. Ε, η έκθεση επιβεβαιώνει ότι δεν έχει αλλάξει η τάση. Πάνω από το μισό, 56% των θυμάτων που καταγράφονται είναι κυρίως γυναίκες και παιδιά. Το 95% έχουν υποστεί ε, σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση. Ε, είμαστε γνώμονες προς τους συναδέλφους της ΛΥΜΠΕ που το αναγνωρίζουν και συνεργάζονται μαζί μας για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, θέλω να δώσω το λόγο στην κυρία Βασιλιάδου, συντονίστρια, για να μας παρουσιάσει τη μελέτη. Και μετά θα ακούσουμε μια αλλαγή απόψεων με τους βουλευτές. Παρακαλώ. Thank you very much. Good morning. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σε όλους. Ε, καλημέρα και σε όσους είναι εδώ για πρώτη φορά. Ε, αναπομονούμε για τη συνεργασία μας. Ευχαριστώ και τις δύο επιτροπές και τους δύο προέδρους. Ε, η συνεργασία μας για τα θέματα καταπολέμησης της διακίνησης ε, ανάγεται σε πολύ, πολύ μακρινό παρελθόν και σας ευχαριστώ για αυτό. Ανυπομονούσα για τη σημερινή συνάντηση και προετοιμαζόμουν και σκεφτόμουν ότι κάποιοι από εσά γνωρίζουν τη δουλειά τη Επιτροπή μα, κάποιοι ίσω λίγο λιγότερα να γνωρίζουν. Γι' αυτό θα παρουσιάσω το βασικό πλαίσιο των πολιτικών. Το δικό μου, η δική μου εντολή αναλύεται στην οδηγία για την καταπολέμηση τη διακίνηση στο άρθρο 20. Μια μοναδική περίπτωση στον επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσπαθώ να προάγω τον συντονισμό μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και φορέων, κρατικών, οργανώσεων τη κοινωνία των πολιτών, με κυβερνητικέ οργανώσει και να οργανώσω τον στρατηγικό μα σχεδιασμό εντό και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει τα μάλα αυτή τη δουλειά. Και έχω δει να υπάρχει υποστήριξη με όλες τις, από όλες τις επιτροπές και από ολόκληρο το Κοινοβούλιο. Πραγματικά υπήρξε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση της διακίνησης και τώρα θα εξηγήσω ποια είναι τα επόμενα βήματά μας. Αυτό που είναι μοναδικό ως προς την καταπολέμηση της εμπορίας και ενώνει τις δυνάμεις όλων των επιτροπών είναι ότι είναι σοβαρότατο έγκλημα και πολύ κερδοφόρο. Το λένε και οι συνθήκες. Πρέπει να καταπολεμάτε, διότι είναι τέτοια παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντίκειται στο άρθρο 5 της Χάρτας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και αυτό είναι μια μοναδική περίπτωση. Είναι και παραμένει ε, πολιτικός τομέας, μάλλον τομέας καταπολέμησης του εγκλήματος που είναι τομέας προτεραιότητας. Θα μπορούσα να σα αναφέρω δεκάδε χιλιάδε παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων που έχουμε στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Θα μου έπαιρνε δυο συνεδριάσει. Θα σα πω ένα μόνο παράδειγμα. Μια 19χρονη άνεργη ε, έρχεται σε επαφή με έναν από του γνωστού τη από άλλο κάτω μέλο και τη λέει Θε να έρθει να δουλέψει σε ένα καφέ, σε ένα μπαρ στην τάδε μεγάλη πρωτεύουσα, μια μετρόπολη και θα σε βοηθήσουμε να βρεις μακροπρόθεσμα μια άλλη δουλειά. Καλύτερε φίλε από το Λύκειο Πήγε λοιπόν, έδειξε εμπιστοσύνη και πήγε στην άλλη πόλη. Πώς πήγε ως εκεί. Κάποιος άγνωστος βοήθησε για να βρει τα χαρτιά να πάει ταξίδι και φρόντισε τα διαδικαστικά. Όμως την κλείδωσαν μόλις έφτασε σε ένα διαμέρισμα Δέκα μήνε έμεινε κλεισμένη εκεί και την υποχρέωσε να παντρευτεί έναν υπήκο τρίτη χώρα, παρέχοντα σεξουαλικέ υπηρεσίε με το ζόρι, διάστηκε στην ουσία, κάτω εξακολούθηση από πελάτε, χρήστε, κακοποιητέ, να του πω έτσι, ε, Ευρωπαίου και μη. Επειδή η αστυνομία σε αυτό το τομέα είναι πολύ καλά εκπαιδευμένη και οι γείτονε το πήραν χαμπάρι, ειδοποίησαν την αστυνομία Ευτυχώς η αστυνομία παρενέβη και την διέσωσε. Ήταν καλό το τέλος της ιστορίας. Εγώ τη συνάντησα σε ένα καταφύγιο για θύματα. Είδα ότι έχει και καρκίνο στους λεμφαδένες και για λόγους που τώρα δεν μπορώ να εκθέσω δεν είχε πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες. Επίσης δεν ήθελε να καταθέσει κατά των διακινητών διότι ήδη την είχαν απειλήσει ότι θα σκοτώσουν τα μέλη τη οικογένειά τη. Ε, το καταφύγιο, επειδή δεν είχε αρκετού πόρου, μπορούσε να την κρατήσει μόνο για ένα δίμηνο. Μετά το πέρα του διμήνου, έμενε άστεγη. Άστεγη, καρκινοπαθή, 19 ετών. Δεν το λέω για να κλάψετε, ή να βουρκώσετε και να αισθανθείτε ικτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για έναν αριθμό νεαρών γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ε, συντονισμένο να αντιμετωπίσουμε αυτές τις περιπτώσεις. Πού πήγαν όλα αυτά τα χρήματα του οργανωμένου εγκλήματος σε αυτές τις ε, συναλλαγές από όταν αυτή η κοπέλα έφυγε από το χωριό της μέχρι να κάνει όλη αυτή τη διαδρομή και να επιστρέψει τελικά πίσω στη χώρα τη. Πού πήγε όλο αυτό το χρήμα που διακινήθηκε σε αυτή την αλυσίδα, δεν έχουμε κανένα ίχνο. Ήταν ε, ε, κάποιο υπεύθυνο ε, από τη μετανάστευση, από τη δικαιοσύνη. Δεν έχουμε κάποιο ίχνο ούτε εκεί. Έχουμε λοιπόν μια περίπτωση παραβίαση τόσων κανόνων και δικαιωμάτων. Είναι στο επίκεντρο της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και είναι τόσοι τομείς που ε, μπλέκονται εδώ σε τέτοιες περιπτώσεις. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα του τι κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε ένα φιλόδοξο νομικό εργαλείο της Ένωσης, πολύ φιλόδοξο, ε, χάρη και στο Κοινοβούλιο και την παρέμβασή σας. Και τώρα κοιτάζουμε τα μέτρα, υλοποιη... Ε, τα μέτρα μεταφοράς στην Εθνική Νομοθεσία. Έχουμε τρει προτεραιότητε και το λέει και η τελευταία ανακοινώση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα να αντιμετωπίσουμε την ε, νοοτροπία αυτή τη ατιμορρησία. Ένα ερώτημα που διαρκώ ανακύπτει, θα το ρωτήσετε σίγουρα, αλλά το απαντάω ε, ήδη από τώρα. Τι έγινε με αυτού του εκατοντάδε άνδρες αυτή την περίπτωση που επισκέφτηκαν αυτή την κοπέλα και την βίασαν στο διαμέρισμα. Η απάντηση είναι ήδη έτοιμη. Τίποτα. Πρέπει αυτή τη συνήθεια τη ατιμορρησία να την αντιμετωπίσουμε για να καταστρέψουμε το επιχειρησιακό μοντέλο τη διακίνηση. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι τα θύματα έχουν δικαιώματα και μπορούν να τα ασκήσουν. Έχουμε πολύ καλό νομικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα των θυμάτων. Πρόσβαση δεν δίνουμε. Πρόσβαση για την άσκηση των δικαιωμάτων των θυμάτων. Εκεί <clears throat> πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Επίση, χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια για την απάντησή μα, την πάταξη τέτοιων εγκλημάτων. Και επίση πρέπει να συντονίσουμε καλύτερα και τη χρηματοδότηση. Σε μια τέτοια υπόθεση έχουμε ένα φαινόμενο που αφορά τη διάσταση των φύλων. Ε, έχει να κάνει με δικαιώματα παιδιών και παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε πολλά νομοθετικά και πολιτικά εργαλεία μα αναφέρονται αυτά. Είναι εγγεγραμμένα. Έχουμε στρατηγική. Έχουμε 40 δράσει που έχουμε υλοποιήσει παρόλα αυτά. Έχουμε μια έκθεση υλοποίηση που μα λέει που έχουν φτάσει τα κράτη-μέλη. Τώρα κοιτάζουμε τα επόμενα βήματα. Δεν θα διστάσουμε να αναλάβουμε οποιοδήποτε μέτρο χρειαστεί εντό του πλαισίου αρμοδιοτήτων τη Επιτροπή. Έχουμε την έκθεση για την εμπειρία των χρηστών και το τι διδάγματα έχουν αντλήσει από τι εμπειρίε των ίδιων των θυμάτων τη διακίνηση. Έχουμε τη δεύτερη έκθεση πρόοδο που θα δημοσιευτεί σύντομα, ε, οργανώθηκε υπό τη δική μου αγίδα, Έχουμε διαδικασίε συλλογή δεδομένων και έχουμε και μια σωρία εκθέσεων για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. Έχουμε πολυάριθμες μελέτες, ένα σωρό δημοσιεύσεις που μπορείτε να τις βρείτε στον στο τοπό μας. Και πάλι θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο, γιατί κάθε φορά που υπάρχει μια δημοσίευση, το Κοινοβούλιο μας προσκαλεί, τη συζητούμε, οργανώνουμε ακροάσεις, διασκέψεις, εργαστήρια και αυτό βεβαίως βοηθά τη διάδοση ε, ε, των, σωστών αρχών και της πολιτική, των πολιτικών μας στόχων. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε με την ε, διακίνηση δεν μας ενδιαφέρει τι θα ήταν καλύτερο ή χειρότερο, μας ενδιαφέρει να το πατάξουμε το φαινόμενο αυτό. Έχουμε λοιπόν ένα δίκτυο υπαλλήλων από όλα τα κρατη μέλη και από ανεξάρτητους φορείς που συναντιόνται δις ετησίω. Εγώ συντονίζω το δίκτυο αυτό σε συνδυασμό ε, με, του, με τις κυλιόμενες προεδρίες του Συμβουλίου. Έχουμε μια επόμενη συνάντηση το Δεκέμβριο υπό την αιγίδα της Συνδικής Προεδρίας και αυτό που είναι μοναδικό είναι ότι έχουμε και μια πλατφόρμα των πολιτών, 100 μη κυβερνητικέ οργανώσεις που λένε ότι αισθάνονται πλέον σαν οικογένεια ε, για την καταπολέμηση της διακίνησης. Συμμετοχή πάρα πολλών ανθρώπων, τεράστιο ευρωπαϊκό δίκτυο, συναντιόμαστε όλοι εδώ και πέντε χρόνια δις ετησίως και πραγματικά έχουν πολύ στενούς δεσμούς όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι συνεργάτε. Αυτό που κάνουμε δις ετησίω, στην αρχή δεν το βλέπαν όλοι πολύ καλά, αλλά τώρα το βλέπουν πιο θετικά. Συνδυάζουμε εκπροσώπου ε, των κρατών μελών με εκπροσώπου τη κοινωνία των πολιτών. Του φέρνουμε στην ίδια αίθουσα να συζητήσουν. Δεν ήταν κάτι που ήταν συνηθισμένο στην κουλτούρα των θεσμικών οργάνων. Η εκπρόσωποι τη κοινωνία των πολιτών θεωρούν ότι ο εθνικό εισηγητή από ένα κάτω μέλο ε, βρίσκεται απομονωμένο στην πρωτεύουσά του και μια μικρή κυβερνητική οργάνωση εργάζεται σε διαφορετική γεωγραφική περιοχή εντελώ. Σε αυτήν την συνάντηση έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στην ίδια αίθουσα και να συνομιλήσουν. Επίση, έχουμε 10 ευρωπαϊκού φορεί από το 2011 συγκεκριμένα. Μοναδική διοργάνωση. Και 10 οργανώσεις θα τις έχετε συναντήσει ήδη σε διάφορες ακροάσεις, που έρχονται για να συζητήσουμε και για το θέμα της αντιμετώπισης της διακίνησης. Η Σέπολη, η ΑΕΓΕ, η ΦΡΑ, η Γιουλίζα και ούτω καθεξής. Τι ξέρουμε τώρα. Την κορυφή του παγόβουνου βάσει της έκθεσης. 30.000 και θύματα μόνο το 2016. Είναι ο πραγματικός αριθμό αυτός. Όχι. Είναι ο αριθμό των θυμάτων που έχουν εντοπιστεί από τις αρχές. Που έκαναν καταγγελία, μήνυση, ε, έφτασαν στο γνωστικό πεδίο τη Επιτροπής. Δεν ξέρουμε του πραγματικούς αριθμού γνωρίζουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων είναι θύματα περιπτώσεων σεξουαλική εκμετάλλευσης κυρίως. Έχουμε όμω και εργασιακή εκμετάλλευση ε, ή την διακίνηση οργάνων που έχουν αφαιρεθεί, καταναγκαστικούς γάμους ή ε, καταναγκαστική συμμετοχή σε οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να εντοπίσουμε θύμα που μπορεί να είναι παιδί. Κάποιες φορές μιλάμε για ε, βρέφη και κάποιες φορές μιλάμε και για 7 χρόνια. Από το 2013 γνωρίζουμε και έχουμε εντοπίσει ότι πολύ συχνά η διακίνηση στρέφεται κατά των γυναικών. Υπάρχει μια γενικευμένη τάση να μετατοπίσουμε το επικεντρό της προσοχής μας από τη σεξουαλική εκμετάλλευση σε κάτι άλλο. Κάποιοι μιλάνε για κόποση. Εάν οι πολιτικοί ηθήνοντες και οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων κουράστηκαν να ασχολούνται με το θέμα. ας τους ζητήσουμε να κάνουν ένα διάλειμμα πριν να ασχοληθούν με την κόπωσή τους. Εγώ θέλω να σας ζητήσω τη σεξουαλική μετάλλευση να τη στο πρώτο. Ε, πρώτη προτεραιότητα τη πολιτική σα δουλειά. Εάν υπάρχει αν υπάρχουν άλλε προτεραιότητε, αν υπάρχει κόπο, αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παραμελούμε την σεξουαλική εκμετάλλευση. Έχουμε μια σειρά από δημοσιεύσει στο σχετικό ιστότοπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορείτε να τι δείτε. Και αυτό που θέλω να τονίσω πάλι σήμερα είναι ότι τα μισά των θυμάτων τη διακίνηση που έχουμε εντοπίσει είναι ε, πολίτε υπηκόοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω, πολλά από αυτά έχουν σχέση και με την μετανάστευση. Βεβαίω, πολλά από τα θύματα είναι μη Ευρωπαϊκή εθνικότητα. Αλλά δεν έχουμε καμία νομική ή ηθική ε, ε, έγκριση και αρχή, κύρος, για να δημιουργήσουμε μια ιεράρχηση, να προβλέψουμε μια ιεράρχηση των θυμάτων βάσει τη εθνικότητα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι λιγότερο θύματα όσοι είναι από τρίτη χώρα. Και σα ρωτώ, τι να πω για αυτή την κοπέλα, αυτή την νεαρή που σα ε, παρουσίασα προηγουμένω. Είναι μια άλλη που γνώρισα σε ένα άλλο κρατός ήταν 13 και είχε και παιδί. Είτε είναι πολίτε τη Ένωση είτε όχι, πρέπει όλου να του προστατεύουμε. Είναι λοιπόν ε, ένα περίπλοκο έγκλημα. Πρέπει να επικεντρωθούμε στην αντιμετώπιση των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ναι, αλλά είναι σοβαρό και ιδιαίτερα κερδοφόρο έγκλημα, εγκληματική δραστηριότητα. Το κέρδο το αποσπούν οι εγκληματίε διακινητέ, έμποροι, αλλά και σε άλλου τομεί που λειτουργούν, μάλλον νόμιμου Φορεί που μπορεί να είναι εμπλεγμένοι σε παράνομες δραστηριότητε. Σε ένα λεωφορείο με 20 κορίτσια που πάνε από το σημείο Α στο σημείο Β χωρίς ένα συνοδό. Είναι ένα παράνομο λεωφορείο φαντάζομαι, με παράνομη άδεια κυκλοφορία. Τι συμβαίνει εκεί μέσα. Πού κοιμούνται, πού τρώνε. Τι είναι αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε, να μάθουμε και θα έπρεπε να γνωρίζουμε. Πού πάνε τα λεφτά, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι καθαρό και εξάστερο. Η διακίνηση δεν συμβαίνει γιατί ο κόσμο έχει προβλήματα, είναι ευάλωτο. Ναι, υπάρχει ανισότητα στη διάσταση στα φύλλα. Ναι, υπάρχει φτώχεια. Ένα βουλευτή πριν από κάποια χρόνια μου είπε: Δεν θα καταφέρετε τίποτα αν δεν ε, κρυζώσετε τη φτώχεια. Εάν έτσι σκεφτόμαστε, δεν θα κάνουμε τίποτα. Η εμπορία, η διακίνηση έχει δύο γενέσφαιρου αίτια. Πρώτον, γιατί κάποιοι βγάζουν ε, μεγάλο, μεγάλα, καταφέρνουν να βγάλουν μεγάλο κέρδο από όλη αυτή τη δουλειά. 30 δις ετησίως υπολογίζεται. Η κορυφή του παγόβουνου μόνο, για τους παράνομού και μόνο, και που πάει αυτό το χρήμα. Και το δεύτερο είναι ότι κάποιο έχει τη διάθεση να εκμεταλλευτεί ένα θύμα. Την νεαρή που σα είπα προηγουμένω. Σκεφτείτε τι. Ήταν πολύ ευάλωτη αν αφαιρέσει κανείς το κέρδος, το παράνομο κέρδος και τους αυτούργους, καταργείται η εμπορία για η διακίνηση. Έχουμε έναν ευάλωτο άνθρωπο που χρειάζεται προστασία και ασφάλεια, αλλά καμία διακίνηση. Αυτή είναι λοιπόν η δική μας τοποθέτηση. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε τηρώντας τα διεθνή πρότυπα. Πρόσφατα κάποιοι άρχισαν να λένε ότι ότι το πρωτόκολλο του Παλέρμο και η, η σύμβαση της Γιούνρα ε, πρέπει να αναθεωρηθούν. Όχι. Δεν χρειαζόμαστε νέα νομικά εργαλεία. Μπορεί να μείνουμε καλοί υπάλληλοι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά όχι. Χρειάζεται η υλοποίηση αυτών που έχουμε σε πρώτη φάση. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε την καταπολέμηση κάθε μορφή εκμετάλλευση. Και σε διεθνέ επίπεδο θα κοιτάμε όλου του βιώσιμου στόχου τη χιλιετία για την αντιμετώπιση τη εμπορία διότι προ στιγμήν ε, ε, ασχολούμαστε μόνο με ένα κάθε φορά με μεμονωμένα και πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όλοι οι τομεί αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ε, κουλτούρα αυτή, την συνήθεια τη ατιμορρησία. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε άλλο αυτό. Τα κράτη-μέλη έχουν κάνει κάποια πράγματα, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχουν κάνει τίποτα και τα λέει και η έκθεση. Αλλά θέλω να κλείσω με το εξή. Έχουμε μπροστά μα, κυρίε και κύριοι, τη μόνη μορφή εγκλήματο που γνωρίζω εγώ και γνωρίζουν και οι ε, υπεύθυνοι δικαστικοί, όπου κάποιο μπορεί εν γνώση του να εμπλακεί εκμεταλλευόμενο άλλου, χρησιμοποιώντα τι υπηρεσίε του, εδώ μιλάμε για βιασμού, αλλά τέλο πάντων, και να μην υπάρχουν και κυρώσει για το συγκεκριμένο έγκλημα. Ενώ η οδηγία το ζητά, ζητά την επιβολή κυρώσεων και τιμωρία, το ζητά από τα κράτη-μέλη να το προβλέψουν, υπάρχουν ακόμα αντιστάσει να ολοκληρώσω. Η έκθεση της Europol. Δείχνουμε σεβασμό για τις εκθέσεις της Europol, για τη διακίνηση των παιδιών. Η εκπόρνευση των ανηλίκων μπορεί να είναι πολύ κερδοφόρα για τους εμπόρους. Οι πελάτες είναι επιρρεπεί στο να πληρώσουν για σεξουαλική επαφή με παιδί συχνά ε, πρέπει να φτάσουν ένα όριο καθημερινά ε, για την υπηρεσία αυτή και για να καλύψουν τα έξοδα στέγασης ή ε, των αντικειμένων εκμετάλλευση. Για παιδιά, 11 χρονών, κορίτσια, ε, πολλές φορές υπάρχουν ομάδες που στοχεύουν συγκεκριμένα παρθένα κορίτσια γιατί πληρώνουν περισσότερο οι πελάτες. Οι πελάτες άμα τους ρωτήσεις λένε δεν το ξέρανε τα εικαζόμενα θύματα διακίνησης που είχε εντοπίσει ο IOM το 2016 από την Ιγυρία, διακινήθηκαν προς την Ιταλία και όλη την Ευρώπη, ε, σα ρωτώ το εξή. Από του αυτούργου και του δράστε που πήραν μέρο στην, εκμετα... στην παράνομη τη δραστηριότητα, στην εκμετάλλευση, ποιοι προσήχθησαν στα δικαστήρια, ποιοι διώχθησαν. Κανένα, μηδέν. Πρέπει λοιπόν αυτό να το σκεφτούμε. Υπάρχουν φοβερά κενά, νομικά κενά, στο πολιτικό μα πλαίσιο. Βεβαίως ασκούμε διώξει στους ε, εργοδότες που ε, εκμεταλλεύονται εργαζόμενους ε, γυναίκες ή παιδιά είτε είναι υπήκοτροι τρίτη χώρα είτε όχι. Αλλά πρέπει να πω το εξή. Είμαι αρκετά μεγάλη για να μπορώ να συζητήσω για θέματα βιασμού και θυμάμαι κάποιου καιρού που ο βιασμό δεν μπορούσε να θεωρηθεί εγκληματική δραστηριότητα. Γιατί έλεγε κανεί πώ αποδεικνύεται. Πού να το ξέρει ότι έγινε. Αυτά είχα να πω εδώ. Πρέπει να πω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θεματοφύλακα των συνθηκών. Παρακολουθούμε την ε, υλοποίηση των ε, μέτρων και των αρχών προβλέπει η οδηγία τα ελέγχουμε. Πρέπει όμω να επικεντρωθούμε στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Πρέπει να τη φέρουμε στο επίκεντρο, ενώ την έχουμε παραγωνίσει τόσο καιρό. Πρέπει να υπάρχει πλέον νομική σαφήνεια. Και πρέπει να σταματήσουμε να κοιτάζουμε να είμαστε μοδάτοι με όρου που δεν έχουν καμιά νομική αξία. Τι θα πει σύγχρονη δουλεία, εξακαναγκαστική, καταναγκαστική εργασία, παιδική εκμετάλλευση, όλα στο ίδιο καλάθι. Όχι. Αυτή είναι μια συνταγή για να αφήνουμε τα θύματα βοήθητα. Τα χάνουμε Πρέπει να πάψει αυτή η συνήθεια τη ατιμορρησία, την κουλτούρα τη ατιμορρησία. Αν σα νοιάζει τι γίνεται με τα θύματα, πάψτε ε, να μην ε, αντιμετωπίζετε του ε, αυτοργού. Αν πάω πάλι πίσω σε αυτή την αιρή γυναίκα που σα είπα προηγουμένω, το πρώτο που λέει είναι θα ήθελα όλοι να πεθάνουν. Εγώ δεν λέω να πεθάνουν, αλλά θα ήθελα να προσεχθούν. Να προσεχθούν σε ένα δικαστήριο με τον τρόπο που προβλέπει ο νόμο. Είναι ο καλύτερο τρόπο να αντιμετωπιστεί και να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα θύματα. Κλείνω λέγοντα ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον νόμο και να τον εφαρμόσουμε επιτέλου. Είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και πραγματικά υπολογίζω σε εσά για να το πράξουμε. Ευχαριστώ κυρία Βασιλιάδου και για το πάθο σα και για τη στράτευσή σα. Και να είστε βέβαιοι ότι τα συμμεριζόμαστε και τα δύο. Εξού και η συνεδρίαση αυτή. συνήθω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ε, αυτά τα θέματα συμβαίνει να απασχολούν και να ενδιαφέρουν πάνω από μία επιτροπή στο Κοινοβούλιο. Βέβαια και την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, όπως έχετε ζήσει και εσείς όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς είμαστε αρμόδιοι για την πολιτική και την νομοθεσία ε, ως προς το ποινικό δίκαιο για να απαντήσει στην εγκληματική διάσταση του τράφικινγκ, αλλά έχει και μια διάσταση φύλου αυτό και το τονίσατε εσείς με πολύ μεγάλη σαφήνεια έχει να κάνει με δικαιώματα των γυναικών, γυναική εκμετάλλευση, ε, ισότητα παντού στην Ένωση. Εδώ λοιπόν έχουμε έδαφος για συζήτηση και μακρύ κατάλογο, αλλά περιορισμένο χρόνο. Θα πάρετε όλοι το λόγο, αλλά παρακαλώ να περιοριστείτε στο ένα λεπτό για να μιλήσουν όλοι. Και να απαντήσει και η κυρία Βασιλιάδου. Ο κύριος Λέναρς, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Εντυπωσιακά αυτά που μας είπατε, κυρία Βασιλιάδου. Είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς σε ένα λεπτό, γιατί είπατε τόσα λεπτά, και, ε, τόσα πολλά και τόσα πολύτιμα. Πολύ σύντομα. Ναι, η οδηγία του 2011 χρειάζεται ε, πλήρη μεταφορά, εφαρμογή και υλοποίηση από όλου τους ενδιαφερομένους. Αυτό δεν το συνειδητοποιούμε τώρα, το ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια. Όταν μιλήσαμε για τη διάσταση του φύλου που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, αυτό το ξέρουμε χρόνια ολόκληρα. Η προστασία των παιδιών, όταν συζητούμε για αυτή, για την ταυτοποίηση και προστασία των θυμάτων. Χρόνια ολόκληρα τα λέμε αυτά, αλλά για κάποιο λόγο ακόμα καθυστερεί και υστερεί η ε, εφαρμογή. Τι πρέπει να γίνει για να γίνεται σωστά αυτή. Μετά, μπορεί ε, να βελτιωθεί κάτι στην αρχική οδηγία, γιατί έχουν περάσει και 8 χρόνια. Δεύτερον, αυτό το έγκλημα ε, συνεχώς εξελίσσεται, αλλάζει. Τον Δεκέμβριο του 2018 σε μια έκθεση μιλήσαμε για στοιχεία του 15 και του 2016. Μήπως πρέπει να βρούμε ένα νέο τρόπο να συλλέγουμε στοιχεία έτσι ώστε οι απαντήσεις μας να είναι πιο κοντά χρονικά σε όσα συμβαίνουν και πιο ευθυγραμμισμένα με τις εξελίξεις. Και τρίτον, ε, ε, εκτιμώ πολύ τη συνεργασία. Αναφερθήκατε στους οργανισμούς και με τις επιθεωρήσεις εργασίας και τις κοινωνικές επιθεωρήσεις. Ελπίζω σύντομα να δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, η ΕΛΕΗ, μπορεί να συνεργαστεί για την αντιμετώπιση τέτοιων ε, καταχρήσεων. Ε, από τους σοσιαλιστές η κυρία Σπούρεκ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ για την καταπληκτική παρουσίαση τα στοιχεία για το 2015-2016 από τη δεύτερη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι οι πέντε πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, καταγεγραμμένων θυμάτων ήταν Ρουμανία, Ουγγαρία, κάτω χώρες, Πολωνία και Βουλγαρία. Αυτές οι χώρες είναι οι ίδιες με το 2010-2012 στην πρώτη έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλύσει για ποιο λόγο αυτές οι χώρες εξακολουθούν να έχουν τις ίδιες στατιστικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Προκατσίνη από το ECR. Grazie. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' Η διακίνηση ανθρώπων είναι το βασικό λόγο για τον οποίο εξακολουθούμε να στηρίζουμε ότι είναι παράλογη η πολιτική ανοιχτών λιμένων για όλους. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε πως πρέπει να προλαμβάνονται οι αναχωρήσεις, να παρεμβαίνουμε για την αντιμετώπιση των αιτίων για τα οποία ε, διαφεύγουν οι γυναίκες από, ε, από τα κράτη τους. Ε, μόλις χτες η Ιταλική αστυνομία εξάρθρωσε με μια οργάνωση που εκμεταλλευόταν τις νικηριανές γυναίκες που κατά χιλιάδες αποβιβάζονται από σκάφη συχνά και των ΜΚΟ στην Ιταλία μπαίνουν σε ένα σύστημα υποδοχής ε, το οποίο προφανώς λειτουργεί, εκμεταλλεύονται το χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους για την ε, ε, διεθνή, διεθνή προστασία και γίνονται εμπόρευμα για τους διακινητές σάρκας και σεξ. Σας ευχαριστώ κύριε Μορκατσίνη. Εσείς δεν, είχατε το, δεν ήσασταν στον κατάλογο, έχετε το λόγο κύριε Εντεφέλτ, εξ ονόματος της, του Renew Europe. Εμένα με τρομοκρατεί η προηγούμενη παρέμβαση που στην ουσία ε, λέει ότι οι γυναίκες είναι οι, οι ένοχες και αυτές που διαπράττουν το έγκλημα ενώ εφόσον έχουν γίνει εμπορεύματα, όπως είπατε προηγούμενο ομιλητέ, σημαίνει ότι υπάρχει αγορά ανδρών οι οποίοι ε, καταχρώνται και κακομεταχειρίζονται αυτές τις γυναίκες. Ακόμα και άνθρωποι σε πολύ ψηλέ θέσεις και πολιτικοί ηγέτες διαφορών χωρών κατηγορούνται για οργάνωση ε, ε, πάρτι οργείων με ανήλικα κορίτσια και θύματα. Ε, εγώ συμφωνώ με τα όσα είπαν οι εκπρόσωποι του ΕΛΚ. Εφαρμογή. Εφαρμογή, γιατί όλοι έχουμε σοκαριστεί και εντυπωσιαστεί και θλιβεί με τα όσα μας είπατε, αλλά όλα οδηγούν στην ίδια, στην ίδια παρατήρηση. Εφαρμογή της νομοθεσίας, όταν ξέρουμε πόσο φρικτά είναι όλα αυτά, ποιο είναι το εμπόδιο. Γιατί εγώ ως ε, βουλευτής θέλω πάντα να ξέρω τι ενέργειες θα κάνουμε για να αντιμετωπιστεί. Ευχαριστούμε κυρία Ιντβέλ, κυρία Μπιόρκ Κουέ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και για αυτή την ε, έκθεση σήμερα. Σας διαβεβαιώ πως δεν υπάρχει εδώ κόποση. Υπάρχουν ε, ε, εκμεταλλευτές και διακινητές γυναικών στην πορνεία, αλλά έχουμε πολιτικές διαφορές και βεβαίως πρέπει να δούμε καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας. Αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να δούμε. Πρέπει να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες, να δούμε ότι τα, τα ε, καταφύγια και οι ξενώνες για τις γυναίκες είναι πραγματικά εξοπλισμένοι και αρκετοί και πρέπει να στάσουμε αυτή την ζήτηση. Υπάρχει ζήτηση, άρα λεφτά αυτοί που εκμεταλλεύονται οι χώρες που δεν έχουν τέτοια νομοθεσία θα πρέπει να σταματήσουν ε, την ζήτηση γυναικών, πορνών. Ε, διαφορετικά θα υπάρχει και συνέχεια το πρόβλημα και κάποιοι προσπαθούν αυτοί να το κάνουν θέμα μετανάστευσης. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να χρησιμοποιούμε αυτό το τομέα πολιτικής ως ένα εργαλείο για να κλείνουμε τα σύνορα της Ευρώπης όπως κάνουν ορισμένοι. Όχι, θα πρέπει να κλείσουμε τα πορνεία, όχι τα σύνορα. Έχουμε δουλειά μπροστά μας και ε, ως αρχή τουλάχιστον να ποινικοποιηθεί η αγορά υπηρεσιών γυναικών που έχουν πέσει θύματα διακίνησης. Να ποινικοποιηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Άντερσον έχει το λόγο. Yes, good morning. And, uh, thank you for the report. Uh, Καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την έκθεση. Α, και τώρα αποφάσισα να μιλήσω γερμανικά ξαφνικά. Ε, η έκθεση είναι εκτενέστατη. Έχουν μερικά ερωτηματικά ανακύψει για μένα. Πρώτο ερώτημα. Τα θύματα, υποτιθέμενα θύματα από πού προέρχονται. Δεύτερον, οι γυναίκες λέτε ε, είναι θύματα αυτής της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλαβαίνει το πρόβλημα ότι έχουμε όλο και περισσότερο δράστες από τις βορειοευρωπαϊκές χώρες που ε, δουλεύουν εκεί στην πορνεία, ας πούμε η Νιγηριανή μαφία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, θεωρεί ότι φταίει ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων, για να μην πω ανύπαρκτος έλεγχος των εξωτερικών συνόρων, που όχι απλώς διευκολύνει το τράφικινγκ, αλλά και το καθιστά δυνατό κατά πρώτο λόγο. Ε, επίσης ε, θέλω να αφαιρθώ σε αυτή την περίπτωση στο Ρόδραμ ε, αν δεν καταλάβατε τι έγινε, ε, πάνω από χίλια παιδιά από διάφορες συμμορίες εκπονεύτηκαν αναγκαστικά. Εσείς τι θα κάνετε γι' αυτό, για τα παιδιά που τα βγάζουν στην πορνεία και τα εκμεταλλεύονται, να μην ξαναγίνονται θύματα όταν δεν τα πιστεύει κανείς ή δεν, δεν τους ακούν οι αρχές. Τελειώνετε και σκεφτείτε και τους υπολείπους, λέει η Πρόεδρος. Συγγνώμη. Ένα λεπτό έχετε. Αν μιλήσετε περισσότερο δεν θα μπορέσουν οι άλλοι να μιλήσουν. Καλώς. Τελειώνω. Πώς προτίθεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει. Τελειώσατε, όχι τελειώνετε. Ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο σας και να σκέφτεστε και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Η κυρία Τζιπόν από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Δεν θα έλεγα εντυπωσιακή, αλλά με πολύ πάθος. Ε, ε, λέγεται ε, ότι γνωρίζουν για τα δικαιώματά τους, αλλά δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά. Στη Γερμανία Έχουμε καλή εμπειρία ε, με μια τηλεφωνική γραμμή για τη βία που μπορούν να αποταθούν τα θύματα ε, που δεν μπορεί κανείς να βρει ούτε τη διεύθυνση IP γιατί είναι κρυμμένη, ούτε να καταλάβουν από πού τηλεφωνεί κάποιος. Αυτό μπορεί να μεταφερθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να επιβληθεί έτσι κάπως πιο έντονα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, η πράσινη, η κυρία Στρίκ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να μιλήσω μαζί των Πρασίνων. Θα ήθελα να σας συγχαρώ, ε, κυρία Βασιλιάδου, για την ομιλία αυτή ε, και για την αφοσίωση και την επιμονή, γιατί πραγματικά το θέμα είναι πολύ περίπλοκο και δύσκολο ε, ε, να καταπολεμήσει κανείς και να το έχει στην ημερήσια διάταξη. Μιλήσατε για τη σημασία της μη ατιμορρησίας. Συμφωνώ απολύτως και το υπογραμμίζω. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να αποφεύγουμε να τιμωρούνται τα θύματα. Γιατί φοβούνται πάρα πολύ να πάνε στην αστυνομία και να μοιραστούν την εμπειρία τους, γιατί λένε θα βρω τον πελά μου. Και επίσης, ιδιαίτερα όταν δεν έχουν χαρτιά και αυτό ισχύει για πολίτες και τρίτων χωρών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως έχει έρθει η ώρα να βεβαιωθούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τους εγγυηθεί δικαίωμα παραμονής εφόσον είναι ε, θύματα του τράφικινγκ για να αισθάνονται ασφαλείς και να μπορούν να τα καταγγέλουν όλα αυτά στην αστυνομία. Και μήπως θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις ΜΚΟ και άλλες οργανώσεις ε, που ακριβώς ασχολούνται με την στήριξη των θυμάτων και την καταπολέμηση της ποινικοποίηση αυτών των ΜΚΟ. Gracias. Ε, señora tiene usted la palabra. Ε, gracias. Solamente plantear... έχετε το λόγο, κυρία Παλόπ. δύο ερωτήματα. Πρώτον, στην έκθεση εκφράζεται την ε, σα, σας γιατί τα κράτη-μέλη δεν δίνουν στοιχεία. Και επίσης, ε, γίνεται λόγος για δευτερογενή θυματοποίηση ε, με την επιβολή κυρώσεων προς τα θύματα. Η οδηγία όμως δεν ε, αντιμετωπίζει κανένα από αυτά τα δύο θέματα. Στο άρθρο 8 δεν κλείνει η δυνατότητα για τα κράτη-μέλη, δεν απαγορεύεται να επιβάλλουν κυρώσεις στα θύματα. Λέει τα κράτη-μέλη ενθαρρύνονται να μην διώκουν, αλλά δεν τους απαγορεύουν να διώκουν τα θύματα και να τα ε, πηγαίνουν στη δικαιοσύνη και στο άρθρο 5, παράγραφος 2 και 4, επίσης μας κάνει εντύπωση, γιατί λέει το 2 ότι ε, τα νομικά πρόσωπα ε, θα πρέπει να προσέχουν, να επαγρυπνούν. Αλλά τι γίνεται με τους δημόσιους οργανισμούς, τα κράτη και τις δημόσιες αρχές στο σημείο 4. Εξαιρούνται και απαλλάσσονται. Άρα, αθώνονται τα κράτη-μέλη. Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα από το γεννησιμιού της οδηγίας. Παρακαλώ, η κυρία Ιόνς Thank you very much. Um, uh, for your... Ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίασή σας. Πραγματικά μας ε, απελπίζει και πρέπει να καταγράψουμε το γεγονός ότι είναι εκατομμύρια αυτοί που υποφέρουν. Μιλήσατε για το πρόβλημα λοιπόν της υλοποίησης και τα νομικά κενά στο, πλαίσιο, στο νομοθετικό πλαίσιο. Μπορείτε να πείτε περισσότερα τι μπορούμε να κάνουμε για να καλύψουμε τις ελλείψεις και τι δυνατότητες αναθεώρησης της οδηγίας υπάρχουν μια χάραξη καλύτερη στρατηγική για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα που υπάρχουν και την ανάγκη για πρόληψη. Και αν έχετε και χρόνο, πείτε μας κάτι παραπάνω για το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε σχέση με το σύνορο που θα δημιουργηθεί και θα υπάρχει, το νέο διάδρομο, αυτήν την τρύπα που θα υπάρξει, που θα είναι παραθυράκι για εμπορία. Με την κυρία Μωρέτη θα τελειώσουν οι ερωτήσεις και θα έχετε συνέχεια πέντε λεπτά κυρία Βανσιλιάδου για να απαντήσετε. Αλλά επειδή είναι πολύ σημαντικά τα ερωτήματα και το θέμα επίση, πάρα πολύ σημαντικό, αν δεν σας φτάνουν τα πέντε λεπτά, παρακαλώ να στείλετε γραπτό στις απαντήσεις σα για να τις διαβιβάσουμε. Γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπω είπατε και εσείς. Η κυρία Μωρέτη. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω για την ε, τόσο πλούσια παρουσίαση και το τόσο καλό περιεχόμενο. Θέλω να πω στον συνάδελφο Προκατσίνη ότι στην Ιταλία οι λιμένες είναι ανοιχτοί. Ουδέποτε έκλεισαν. Διότι έχουμε διεθνείς συνθήκες και πρέπει να τις εφαστούμε. Και επίσης στην Ιταλία υπάρχει και δικαστικό σύστημα που λειτουργεί ευρυθμότατα και σέβεται τους κανόνες. Τους επιβάλλει μάλιστα και στους πολιτικούς ηθήνοντες. Υπάρχει ένα ζήτημα όμως εδώ με τη Μεσόγειο, ε, διότι και στη Λιβύη ξέρουμε ότι τα πράγματα έχουν φτάσει στο προχώρητο. Υπάρχουν ε, πραγματικά στα τόπεδα συγκέντρωσης στη Λιβύη, όπου βιάζονται οι γυναίκες, Ασχέτως φίλου βέβαια και στους άνδρες υπάρχουν ε, ασκείται σωματική βία και οι άνθρωποι αυτοί απλώς διαφεύγουν. Διαφεύγουν από αυτά τα σε τις φυλακές. Θα έπρεπε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να φροντίσει να μην υπάρχουν τέτοιες συνθήκες, να μην φτάνουν οι άνθρωποι αυτοί να ρισκάρουν τη ζωή τους γιατί δεν μπορούν άλλο να ζήσουν έτσι. Δεν μπορεί να γίνεται παραδεκτό η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανέχεται τέτοιε καταστάσει. Και από εκεί ξεκινάνε και όλα τα προβλήματα που σήμερα συζητάνε βεβαίω. Πρέπει να δούμε το θέμα τη βεβαιότητα τη ποινή σε πρώτη φάση, για ποιον διαπράττει τέτοιου είδου έγκλημα. Και επίση τη δίκαιη, τη νόμιμη και ένομη υποστήριξη των θυμάτων. Στη δική μα την Επιτροπή, την ΦΑΜ, υποβάλαμε ήδη μια νέα φιλόδοξη στρατηγική παρακαλώ, ολοκληρώστε. Για να, εκριζω... να καταργήσουμε, να εξαλείψουμε την εμπορία των ανθρώπων και να ενισχύσουμε την επιβολή ποινών σε όσου εκμεταλλεύονται αυτού του ανθρώπου. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια θετική εξέλιξη εδώ. Ο κύριο Ρομπέρτη, επίση επίσης ε, μου είπαν ότι ζήτησε το λόγο και θα είναι εκείνο ο τελευταίο. Ε, Σα ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω απλά να ευχαριστήσω την κυρία Βασιλιάδου για την ε, εισήγησή του, και για τι πολλές ε, και πολυσχεδείς πληροφορίες που μας έδωσε. Δυστυχώς ενώπιον ενός φαινομένου πλανητικών διαστάσεων, για το οποίο λέγεται ότι ε, πρόκειται για ε, περίπου 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι μπαίνουν μέσα σε αυτά τα κυκλώματα ετησίως και σε σχέση με τις τραγωδίες αυτές που εκτελήσονται, οι έρευνες και το ποινικό στοιχείο το, είναι ακατάλληλο, όχι μόνο στην Ιταλία τη χώρα μου, αλλά σε ολόκληρη την Ένωση. Εφόσον λοιπόν η ποινική διαδικασία, δηλαδή η καταστολή, η καταδίκη των ε, ευεύθυνων για την ε, διακίνηση ανθρώπων δεν αρκεί, γιατί έχει ξεπεραστεί, τότε δεν λειτουργεί και προφανώς η διεθνή συνεργασία. Ε, η διεθνή συνεργασία. Μου λέτε ότι υπάρχουν ε, οργανισμοί που εξασφαλίζουν την κυκλοφορία των πληροφοριών. Εγώ διερωτώ με πώς είναι δυνατόν, ε, εφόσον έχουμε όλες αυτές, όλη αυτή τη μάζα πληροφοριών, οι έρευνες οι αστυνομικές να είναι τόσο ελλειπείς και τόσο σποραδικές. Το πρόβλημα είναι ότι η διεθνή συνεργασία δεν, ε, δεν αρκεί. Ε, για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα στην Ιταλία και αναφέρομαι κυρίως στη διακίνηση ανθρώπων Ολοκληρώστε παρακαλώ διακόπτη η πρόεδρος. Ε, ναι, σε σχέση με την ε, μαφία της Νιγηρίας υπάρχει τώρα ένας Νιγηριανός εισαγγελέα στην Ιταλία που εξασφαλίζει την διασύνδεση ανάμεσα στην Ιταλία και την Νιγηρία. Θα σας πάρω το μικρόφωνο δεν ολοκληρώσετε. Τι γίνεται λοιπόν για να καλυφθεί αυτό το κενό της ελληπούς διεθνούς συνεργασίας. Ευχαριστώ. Η πρόεδρος ευχαριστώ. Και τώρα Συγγνώμη που σας ε, πιέζω, αλλά πρέπει να έχουμε χρόνο για να ακούσουμε και τις απαντήσεις. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ε, ε, ωραία ώρα, ε, γιατί εμένα μου δίνει κίνητρο και όρεξη, το βλέπω, τη βλέπω το ενδιαφέρον σας. Έχω 20 δευτερόλεπτα όμως για να απαντήσω σε κάθε ερώτηση. Εάν δεν σας απαντήσω, να μου το θυμίσετε παρακαλώ και ευχαρίστως θα απαντήσω γραπτός. Πρώτον, για την εφαρμογή της οδηγίας που... Ε, πράγμα που προέκυψε επανειλημμένα. Δεν είχα χρόνο στην εισήγησή μου να πω ότι πρώτα απ' όλα στην έκθεση έχουμε και πολλά θετικά στοιχεία όσον αφορά την εφαρμογή. Έχουμε καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στις αρχές, έχουμε καλύτερη ε, κάλυψη ε, των, θυμάτων, περισσότερο συντονισμό, καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κοινών ομάδων και των οικονομικών ε, ερευνών. Πολλά μέλη, κράτη-μέλη χρησιμοποιούν τη στήριξη των ευρωπαϊκών οργανισμών. Έχουμε δείξει ότι όλο ένα και περισσότερο χρησιμοποιείται η οδηγία. Η ίδια η κοινωνία των πολιτών στη συνεργασία της με τις αρχές έχει βελτιωθεί. Υπάρχουν πολλά πράγματα λοιπόν που πάνε καλά, αλλά ζούμε σε καιρούς και για να το πω ομά, υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη ευαισθησία, πολλά, πολύ ευάλωτοι άνθρωποι και πάρα πολλά κέρδη. Αυτό είναι το θέμα. Ε, ε, πάει πάνω πάνω στη λίστα μαζί με τα όπλα και τα ναρκωτικά. Το να σκεφτείτε ότι είναι τόσο εύκολο να σταματήσουμε τη ροή χρημάτων δεν είναι τόσο εύκολο. Αλλά εγώ παρακαλώ όλους μας θέλω να μας παροτρύνω να ψάξουμε πού βρίσκονται αυτά τα χρήματα και εκεί αυτό θα σημάνει τη διαφορά. Πολλά από τα άρθρα τη οδηγίας εμφαρμόζονται με ενθαρρυντικό τρόπο, αλλά έχουμε χαμηλό αριθμό ε, προσαγωγών και καταδικών. Για, ε, ε, τώρα, για τα στοιχεία. Στοιχεία, ναι, έχουμε από το 16. Ωραία αλλά δημοσιεύουμε τα στοιχεία ταυτόχρονα με το γραφείο του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά και το έγκλημα. Όταν έχουμε να κάνουμε λοιπόν με ποινικέ στατιστικές και δεν θέλουμε έτσι ε, γενικά και αόριστα νούμερα όπως κάνουν κάποιοι διεθνείς οργανισμοί, τότε πρέπει να έρθει σε επαφή με τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες και εγώ πιέζω πολύ ώστε να εξασφαλίσω πως όλοι οι αναμειγνυόμενοι φορεί και η ΜΚΟ και ο ε, θα ε, συμμετέχουν στη σωστή και στην εξασφάλιση της σωστής συλλογής των στοιχείων. Τώρα έχουμε ξεκινήσει την προσπάθεια που θα προκύψει το 2020 για τις τελευταίες στατικιστικές που θα έχουμε. Προσπαθούμε λοιπόν κάθε φορά να βελτιώσουμε την ποιότητα των δεδομένων, αλλά αμφιβάλλω αν μπορούμε να βελτιώσουμε <coughs> και την ταχύτητα με την οποία εκπονούνται οι στατιστικές. Τώρα, εδώ πέντε χρόνια μιλάω για το, στο Ευρωκοινοβούλιο ε, για, για την ανάγκη να κατανοήσουμε και να χρηματοδοτήσουμε περισσότερο το θέμα της ε, διακίνησης για εκμετάλλευση ε, Έχουμε και με την επιθεώρηση εργασίας ε, συνεργασία και αυτό δεν το λέμε περηφάνεια. Το λέω για να σας πω ότι κάνουμε μια μακροχρόνια μελέτη τα τελευταία 15 χρόνια για να δούμε πού πήγαν αυτά τα χρήματα και στη μεγάλη πλειοψηφία τα διπλάσια ήταν στην εκμετάλλευση εργασίας. Για τις χώρες προέλευσης, ναι, εντάξει, ναι, ήρθατε κοντά για να με σταματήσετε σε δύο λεπτά. Μάλιστα, θα σταματήσω. Έχουμε πέντε χώρες το εξηγήσατε. Αλλά να αντιστρέψω το ερώτημα. Από εκεί έρχονται τα θύματα. Αλλά οι εκμεταλλευτές τους είναι εκεί. Εκεί είναι αυτοί που βγάζουν τα πολλά λεφτά. Είναι κοινή ευθύνη λοιπόν. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα να αλλάξω τι, πόσο ευάλωτοι είναι οι άνθρωποι στη Ρουμανία π.χ. Αλλά αυτό που μπορώ να κάνω είναι να δουλέψουμε μαζί, να δούμε όταν φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι, πού πάνε και γιατί. Και νομίζω πως αυτό απαντάει σε διάφορες ερωτήσεις. Θέλω να επαναλάβω. Έχουμε θύματα. Τα μισά είναι ε, υπηκόοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το θέμα των συνόρων και μη συνόρων είναι άσχετο. Είναι, δεν έχει να κάνει. Γιατί τα μισά θύματα είναι υπήκοοι της Ένωσης. Αυτό είναι γεγονός. Και το ένα στα τέσσερα θύματα είναι θύμα η οικογενειακή διακίνηση, μάλλον εγχώρια διακίνηση, δηλαδή στην ίδια του τη χώρα. Να πω στο Βέλγιο, ας πούμε, είναι, ε, είσαι Βέλγος, ο οποίο έχει πέσει θύμα διακίνηση μέσα στο Βέλγιο και δεν πρέπει να με τη, λάθρο τη λαθροδιακίνηση με τη διακίνηση. Ε, το, η λαθροδιακίνηση είναι κατά του κράτους, ενώ η διακίνηση είναι κατά του ίδιου του ατόμου θα μπορούσα να σας πω, ναι, χρειαζόμαστε πολλές νομοθεσίες κατά της διακίνησης ανθρώπων. Αλλά όχι, δεν χρειαζόμαστε. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι να πιέσουμε περισσότερο τα καθημέλια στην να εξασφαλίσουμε ότι ποινικοποιούν αυτούς υπηρεσίες των θυμάτων. Ναι, αυτό πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε ε, σοβαρές... Ε, ε, συντρέχουσες ε, συνθήκες για τους ε, δημόσιους υπάλληλους. Έχουμε μια μοναδική νομοθεσία, το άρθρο 5, που θεωρεί υπόλογες τις νομικές οντότητες, το χρησιμοποιούν τα νομικά πρόσωπα. Αυτό πρέπει να το κάνουμε στα κάτι μέλη. Μιλάμε για πολύ χρήμα, είναι οργανωμένο έγκλημα. Μιλώ για τα θύματα, γιατί αυτούς έχω στην καρδιά μου. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι τα θύματα συνέχεια να λέμε στα θύματα, μα σταματήστε να πέφτετε θύματα διακίνησης. Όχι, τους διακινητές πρέπει να σταματήσουμε, τους πελάτες, ε, τους χρήστες, τους, τους ε, ανθρώπους που χρησιμοποιούν αυτή τις υπηρεσίες. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, αυτούς πρέπει να σταματήσουμε. Και ναι, πρέπει να ακολουθήσουμε τα λεφτά. Γιατί δεν μπορούμε να λέμε ναι, ή ο Νιγηριανός διακινητής και ο Ρουμάνος διακινητής και ο Κύπριος ας πούμε διακινητής, καθώς εγώ είμαι από την Κύπρο. Δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν ένα νέο κορίτσι 7 ετών να φύγει από την Νιγηρία για να έρθει ας πούμε στις Βρυξέλλες μόνο με έναν άνθρωπο δίπλα τη. Είναι ένα σωρό που την πάνε. Λέγοντας ο Τάδε και ο Δίνα είναι υπεύθυνοι, εμείς αποφεύγουμε την ευθύνη που πρέπει εμείς να αναλάβουμε. Είναι μια ολόκληρη αλυσίδα και όπου μπορούμε να τη σταματήσουμε την αλυσίδα, είτε είναι ο οδηγό λεωφορείου, είτε είναι ο υπάλληλο, ο, τύπος στο χωριό της Νιγηρίας, οπουδήποτε και είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Ε, οι γραμμές οι τηλεφωνικές, κάναμε μελάτη, με μια μελέτη. Η πραγματικότητα είναι ότι τα περισσότερα θύματα δεν σκέφτονται καν ότι είναι θύματα ε, διακίνησης. Όχι, λένε, αυτός εκεί με βίασε, εκείνος εκεί με κλείδωσε στην αποθήκη, στο αγρόκτημα. Όχι. Το θέμα είναι να μπορέσει η κοινωνία να χειραφετηθεί, να χρηματοδοτηθεί η κοινωνία των πολιτών, εκεί που αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται. Η άμεση χρηματοδότηση της Κομισιόν έχει αυξηθεί αστρονομικά. Ε, βρίσκουν νέο τρόπος να κάνουν συμμαχία στα κράτη-μέλη. Θα ήταν σπουδαίο να έχουμε μια τέτοια τηλεφωνική γραμμή επίγουσας ανάγκης, αλλά οι μελέτες δείχνουν ότι όχι, δεν είναι αυτός ο τρόπος. Δεν λέω πως δεν θα πρέπει να γίνει σε εθνικό επίπεδο, πάντως όχι σε ευρωπαϊκό. Δεν βοηθάει. Και πολλά ακόμα για την οδηγία και τη ρήτρα περί τιμωρίας. Είναι σαφής και αυστηρή αυτή η ρήτρα. Εγώ νομίζω πως θα πρέπει να την εξετάσουμε και, σε... και μην ξεχνάτε παρακαλώ μια οδηγία αφορά τις μήνυμου προδιαγραφές. Όταν βλέπετε αυτό το φιλόδοξο άρθρο εδώ, είναι ωστόσο μήνυμα προδιαγραφές. Έχω μιλήσει με εισαγγελεί ε, με δικαστές και τα και να ρωτήσω γιατί. Δεν, θέλω να με, δεν είμαι νομικός και δεν θέλω να με, παρα, να με παρανοήσετε, αλλά ας πούμε έχουν δοθεί παραδείγματα για πολύ σοβαρά δικήματα και εγκλήματα και δεν μπορούμε να αποφασίσουμε εκεί το βαθμό στον οποίο θα εφαρμοστεί η ρήτρα μη τιμωρίας. Αν και εκεί πιέζουμε, φυσικά και πιέζουμε. Και για την άδεια παραμονή. Ξέρω πως υπάρχει μεγάλο ε, προβληματισμός, αλλά η οδηγία του 2011 μεταχειρίζεται επί ίσης όλα τα θύματα διακίνησης ανεξάρτητα από το καθεστώς τους. Ήμουν μάλιστα εγώ υπεύθυνη τότε και εκεί έχουμε προσαρτήσει την έκθεση για την οδηγία 2004 που αφορά την άδεια παραμονή. Και ακριβώ λόγω τη ανησυχία μου. Η οδηγία ορίζει συγκεκριμένου κανόνε σε σχέση με τι άδειε παραμονή ε, όσον αφορά υπηκόστη των χωρών, αλλά η οδηγία 11-2011, δηλαδή αυτή περί διακίνησης, ε, ισχύει ως οριζόντιο πλαίσιο ώστε να παρεμποδιστεί η διακίνηση θυμάτων για Ευρωπαίους και μη Ευρωπαίους πολίτες. Τα δύο θα πρέπει από κοινού να αναγνωστούν και να ερμηνευθούν και η εφαρμογή τους θα πρέπει να αξιολογηθεί σαν σύνολο. Υπάρχουν ε, περιπτώσεις όπου έχουν αυτά εφαρμοστεί σωστά και τα είδαμε αυτά στις αναφορές και αυτό θα είναι το, ε, το στόχος, αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να εξεταστούν από κοινού. Πάρα πολλές ερωτήσεις, δεν ξέρω σε πόσες απάντησα. Ναι, νομικά κενά, σημαντική ερώτηση επίσης. Κύριε Γνώμη, κυρία Βασιλιάδου, έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας. Μιλάτε 10 λεπτά. Όχι, όχι, εντάξει, βεβαίω. Ε, κλείστε, κλείστε. Αλλά να το έχετε υπόψη σα, γιατί έχουμε και άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη μέχρι να κλείσουμε το πρωινό. Καλώ. Για τα νομικά κενά. Ε, έχει σημασία και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό έχει χαράξει προτεραιότητες και είναι μεγάλη προτεραιότητα ε, στην ανακοίνωση του 2017 ότι θα πρέπει να εθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να ποινικοποιούν ε, όλοι όσοι γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούν υπηρεσίες θυμάτων. Πάντα το δίνω αυτό το παράδειγμα γιατί δεν το χωράει ο νους μου. Μπορείς να αγοράσεις 30 ευρώ μία τσάντα ε, υποτίθεται designer, μαϊμού και, και σου επιβάλλουν κυρώσεις που καλά κάνουν. Αλλά δεν επιβάλλουν τις ίδιες κυρώσεις όταν χρησιμοποιείς τις υπηρεσίες ενός προσώπου που ξέρεις ότι είναι θύμα και μην μου λέτε τώρα ότι είναι δύσκολο να ε, αποδειχτεί είσαι Νιγηριανή 11 χρονών η η χειμώνα στο δρόμο α δεν το ήξερες α δεν το ήξερε ο άλλος ότι ήταν την άλλη φορά να του με πάρει τηλέφωνο να του το πω εγώ είναι σαν την νομοθεσία για το βιασμό πριν από 20 χρόνια από το 2009 η νομοθεσία λέει όσοι χρησιμοποιούνται όσοι χρησιμοποιούν ε, ως ε, επιχειρηματίες, ως εργοδότες αυτές τις υπηρεσίες δημιουργούνται. Το έχουμε αυτό για την εργατική νομοθεσία για πολίτες τρίτων χωρών. Ενώ εδώ έχουμε νομικό κενό που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ενθαρρύνουμε όλα τα κράτη-μέλη να το κάνουν. Πρέπει να σταματήσουμε τη ροή των χρημάτων και την εκμετάλλευση. Μόνο τότε θα σταματήσει το τράφικινγκ. Και πάμε και βοηθάμε τα θύματα και πίνουμε και το τσαγάκι μας και αισθανόμαστε καλά γιατί βοηθούμε τα θύματα. Για ρωτήστε όμως το γείτονά σας, το παιδί του, ε, τι σημαίνει να τον κλειδώσουν σε μια αποθήκη και δεν βλέπει το φως της ημέρας ε, τρία χρόνια. Και τι, τι αισθάνεται όταν τον σώζουν, υποτίθεται. Ερχόμαστε πολύ αργά. Θα πρέπει να σταματήσουμε αυτή την εκμετάλλευση και αυτή την κουλτούρα και την οτροπία της ατιμορρησίας. Περί αυτού πρόκειται. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βασιλιάδου. Βλέπετε λοιπόν πόσες ερωτήσεις κάναμε. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα αυτά και σαφής η απαντήση σας ότι συμφωνούμε μαζί σας και το λέτε και πολύ ομά και έξω από τα δόντια. Το κοινοβούλιο είναι νομοθέτης και αυτό θέλει ακριβώς να αναγκάσει τα κράτη-μέλη να κάνουν εθνική νομοθεσία γι' αυτό και να προστατεύουν όχι μόνο τα θύματα αναφερθήκατε σε εξωφρενικές περιπτώσεις, δραματικές, ε, με τραγωδίες, αλλά και πώς θα αυξήσουμε την ε, συνειδητοποίηση όλου αυτού του κύκλου ανθρώπινης εκμετάλλευσης. Και μόνο η ύπαρξη της δικής σας θέσης και το πάθος που βάζετε εκεί και η ψυχή που βάζετε πραγματικά είναι πάρα πολύ αξιέπαινα. Θα σας ξαναδούμε σίγουρα γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Και προχωρούμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ε, ε, αποχαιρετούμε τα μέλη της Επιτροπής Γυναικών. Ευχαριστούμε που ήσασταν παρόντες. Το επόμενο θέμα δεν σας πολύ ενδιαφέρει. Έχει να κάνει με ε, τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΒΕ, τα οποία παρακαλώ να παραμείνουν. Και τη χάνει και ο συγκητή σας εκεί. Σας ευχαριστώ. Muchas gracias.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 esta, sórdida dimensión de realidad. Σε ένα τέταρτο θα χάσουμε τους διερμηνείς. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ μεγάλα περιθώρια λιγμό και σας ευχαριστώ που παραμείνατε ε, εδώ τα μέλη της Επιτροπής μας για το τεταρτάκι που μας έχει απομείνει μέχρι να σχολάσουν οι διερμηνείς. Για να μας εγκαταλείψουν. Τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη και την χάνω εγώ εισηγητή σας. Πρόκειται ε, για την εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της σύναψης από τη Eurojust συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Eurojust και της Σερβίας. Γνωρίζετε ότι η Eurojust την περασμένη εβδομάδα κατέθεσε το σχέδιο συμφωνίας. Υπήρξαν και άλλες συμφωνίες με τρίτες χώρες, ε, όπως μεταξύ Αλβανία, Γεωργία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Ουκρανία, Ηνωμένε Πολιτείες, Ελβετία και Μολδαβία. A very short Ε, επειδή ήταν πάρα πολύ ε, σύντομη η προθεσμία, οι ε, συντονιστές συμφώνησαν τον Ιούλιο ε, να ακολουθήσουμε απλουστευμένη διαδικασία. Και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν θα καταθέσουμε τροπολογίες επί της διαδικασίας. Επίσης αποφασίστηκε ε, εγώ ως Πρόεδρος να αναλάβω αυτό το θέμα ως εισηγητής. Θα ήθελα να θυμίσω ότι το Συμβούλιο είχε ζητήσει από το Κοινοβούλιο με επιστολή της 9ης Ιουλίου να γνωμοδοτήσει το συντομότερο και το αργότερο εντός των πολύ τριών μηνών. Στις 11 Ιουλίου συμφώνησαν οι συντονιστές να προχωρήσουν με αυτόν τον τρόπο, λόγω του επίγοντος χαρακτήρα. Αν δεν διαφωνείτε λοιπόν στο σχέδιο έκθεσης που σας υποβάλλω, να θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται. Για να πάει στην Ολομέλεια και να ψηφιστεί τον Οκτώβριο, στην πρώτη Ολομέλεια του Οκτωβρίου. Να ληφθεί η τελική απόφαση για τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω πάρα πολύ σύντομα το σχέδιο έκθεσης. Η Συμφωνία Συνεργασίας Eurojust Σερβίας ακολουθεί ένα μοντέλο αντίστοιχων συμφωνιών που έχει κάνει Eurojust ε, για την ε, δικαστική συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Ε, συμφωνία με τη ΦΥΡΟΜ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Βηγία, με την Ελβετία, Αλβανία και πιο πρόσφατα με τη Γεωργία. Πάντα Eurojust με τις χώρες αυτές. Αυτές οι συμφωνίες μεταξύ άλλων προβλέπουν αξιωματικούς συνδέσμους, σημεία επαφής και ανταλλαγή πληροφοριών σε τακτική τα χρονικά διαστήματα. Η συμφωνία που σας αναφέρω ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Δυτικά Βαλκάνια του 2018. Αυτό ήθελα να το τονίσω επίσης. Άλλες υποψήφιες χώρες προς ένταξη της ε, περιφέρειας εκεί, δηλαδή το Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία, ήδη έχουν συνάψει τέτοιες συμφωνίες. Η Σερβία είναι η τρίτη χώρα, είναι υποψήφια χώρα. Είναι η τρίτη χώρα από πλευράς αιτήσεων συνεργασίας σε αριθμό. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι η χώρα από την οποία ζητούμε περισσότερες προφορίες στην περιοχή και γενικότερα ε, στις περιπτώσεις και τις υποθέσεις που έχει Eurojust, η πιο σπουδαία χώρα. Το 2018 και μόνο συμμετείχε σε, παρακαλώ, 34 υποθέσεις η Σερβία. Άρα ε, δικαιολογείται συμφωνία με τη Eurojust. Στη δεύτερη έκθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε τη σημασία των ομάδων οργανωμένων εγκλήματος όπου συμμετέχουν Σέρβοι πολίτες εξακολουθούν επίσης να είναι από τα πιο συχνά θύματα τράφικινγκ διακίνησης ανθρώπων η Σέρβοι, ε, διακίνηση από τα Δυτικά Βαλκάνια και επίσης υπάρχουν και πάρα πολλά όπλα, απόθεμα όπλων στη Σερβία, το οποίο από μόνο του συνιστά κίνδυνο ε, στα πλαίσια της διακίνησης και του λαθρεμπορίου πυροβολών όπλων. Τέλος, η Σερβία είναι μέρος ε, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Δεδομένων και του συμπληρωματικού πρωτοκόλου. Η ΔΕ Σερβία επίσης ε, ενέκρινε νέα νομοθεσία μόλις το 2018 για την προστασία των δεδομένων. Ε, το κοινό εποπτικό όργανο της Eurojust νομοδότησε θετικά ε, για τις διατάξεις αυτής της συμφωνίας ως προς την προστασία των δεδομένων βάσει όλων αυτών που σας είπα, σας προτείνω να υποστηρίξετε την ε, συμφωνία. Δεν ξέρω αν διαφωνεί κανείς, θέλει να πει κανείς σας τίποτα. Ζητεί κανείς το λόγο. Αλλιώς να θεωρήσουμε ότι εγκρίνεται αυτή η συμφωνία για να περάσει στην Ολομέλεια τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την επίγουσα διαδικασία που ζητήσαμε. Συμφωνείτε με όλα αυτά που σας είπα. Ωραία. Σας ευχαριστώ και τελειώσαμε εγκαίρως. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Επανάληψη συνεδρίασης εδώ στην ίδια αίθουσα το απόγευμα στις 2 η ώρα, μεσημέρι, 2 μετά μεσημβρίας. Το επόμενο θέμα, παρουσίαση των δραστηριοτήτων των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τομέα Δικαιοσύνη και των ιστορικών υποθέσεων. Frontex παρακαλώ. Καλή σας όρεξη.